Bien, και κύριοι, συγγνώμη για την μικρή αυτή καθυστέρηση. Υπήρχαν μερικά τεχνικά προβλήματα που λένε. Είναι φορτωμένη η μερίσια διάταξη με θέματα Αφγανιστάν. Σήμερα δεν θα υπάρχουν δανέζικα, φιλανδικά, σουηδικά, λεπτονικά, σλοβενικά, Μαλτέζικα κλπ. Και σας υπενθυμίζω ότι μόνον τα πλήρη μέλη έχουν δικαίωμα σε διερμηνία. Γι' αυτό. Η συνεδρίαση αναμεταδίδεται και στο web stream. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Λοιπόν, την Τετάρτη στις 6.30 μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών θα δεχθούμε την κυρία Όλι Μπράιντ ως επικεφαλής της ομάδας σοφών που διαπραγματεύεται τη νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ. Φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρεστε πολύ να πάτε την Τετάρτη λοιπόν. Και τώρα το σημερινό μας θέμα το Αφγανιστάν. Στην υποεπιτροπή μας δεν θελήσαμε ούτε και γίνεται να καλύψουμε το σύνολο της κατάστασης του Αφγανιστάν γιατί και στην επέξταση ζητηθεί ευρύτερα. Σήμερα λοιπόν θα περιοριστούμε στην πτυχή που αφορά την ασφάλεια. Τομέα στον οποίο είναι ιδιαίτερα ενεργή η Ένωση οργάνων δηλαδή της αστυνομίας, των δομών του Υπουργείου Εσωτερικών κλπ. Γι' αυτό οι πρώτοι που θα πάρουν το λόγο θα είναι ο κύριος Κλάμπενχάουερ, τον οποίο έχουμε συναντήσει και προηγουμένως, που είναι επικεφαλής των ε, πολιτικών ε, επιχειρήσεων της Ένωσης και μετά θα μας μιλήσει και ο υπεύθυνο της ε, Ευρωπόλ στην Καμπούλ. Θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε συνεχώς ατέρμονες ερωτήσεις, γιατί το θέμα είναι ευρύ βέβαια, αλλά να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Ζήτησα επίσης τον, από τον κύριο Ντέιβις και την κυρία Κατκάρ να έρθουν από την Βεσβία των ΗΠΑ για να μας εξηγήσουν την καινούργια αμερικανική στρατηγική όπως την εξέθεσε ο πρόεδρος Ομπάμα στο West Point και την αμερικανική αντίληψη και κρίση για τις προσπάθειες που γίνονται για την οργάνωση των δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν. Επίσης ο προεδρευτής του Αφγανιστάν θα προσέλθει σε λίγο και μετά θα γίνει και ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Αριάν Καντιέ η οποία μόλις δημοσίευσε ένα βιβλίο για την κατάσταση στο Αφγανιστάν το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα και μας και τον ΝΑΤΟ και την Αφγανική κυβέρνηση. Έτσι θα έχουμε και μια έτσι για να το πω έτσι πιο ανεξάρτητη άποψη. Λοιπόν αυτά για τις παρουσιάσεις και τώρα Έχουμε και τον συνάδελφο της Μπερμάν που είναι μέλος της αντιπροσωπείας με το Αφγανιστάν. Παρακαλώ όλους να είστε σύντομοι και σύντομες γιατί θα μιλήσουν πολύ και γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί η ποιότητα της συζήτησή μας από το αν αποφύγουμε δηλαδή να πλατιάσουμε. Ο κύριος Κλάμπενχάουερ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ντάνσα. Πράγματι είναι δεύτερη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας, στην Υπο-Επιτροπή σας. Την πρώτη φορά όμως έρχομαι εδώ ενώπιον σας βάσει της νέας συνθήκης. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η στιγμή που διανύουμε, διότι επίκειται η διάσκεψη του Λονδίνου και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ενεξελίξη. Θα προσπαθήσω να σας σκιαγραφίσω την κατάσταση μαζί με τον ε, κύριο Βίτρουπ, τον επικεφαλής των ε, αστυνομικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, εδώ και τρία χρόνια διανύουμε μια νέα περίοδο που άρχισε τον Ιούνιο 2007 με κάποια σπουδή. Επρόκειτο για μια αποστολή που είχε πολλά ε, προβλήματα επάνδρωσης, γι' αυτό άργησε να τεθεί σε εφαρμογή μερικούς μήνες. Καταβλήθηκαν όμως μεγάλες προσπάθειες για να τα βάλουμε όλα σε ένα βλάκι και η UPOL έχει μπει σε ένα αυλάκι με τη συφορά του κυρίου Βίτρου. Πρόκειται για έναν βασικό παράγοντα μέσα στα πλαίσια της ε, μεταρρύθμισης του Αφγανιστάν. Η ε, Ιούπολ μπορεί να προβεί σε πραγματογνωμοσύνη ως προς μη στρατιωτικά θέματα. Με βάση αυτή την ε, πραγματογνωμοσύνη και πειρά ο κύριος Άτμαρ, ο οποίος η αποστολή και η... ο τίτλος του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Αφγανικό Κοινοβούλιο είναι επικεφαλής της UPOL ε, και ασχολείται και με την καταπολέμηση του εγκλήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης ε, συνεργάζεται μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς. Είναι από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Έτσι, έχουμε ταχθεί επικεφαλή σε αυτούς τους τομείς. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και η αξιοπιστία μας εξαρτάται από το πώς θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις αυτές. Όταν αποτιμήσουμε τη δράση της UPOL, και αυτό είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οποιαδήποτε μέτρα αφορούν την μεταρρύθμιση των αστυνομικών αρχών με βάση τις δυσμενείς συνθήκες θα πρέπει να ειδωθεί με μια ειδική οπτική γωνία από πλευράς δηλαδή χρόνου εφαρμογής. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια στρατηγική εξόδου. Άρα δεν μιλάμε για στρατιωτικές επιχειρήσεις εδώ, μιλάμε για καθαρά για μια καθαρά πολιτική επιχείρηση. Σε αντίθεση με τον ΝΑΤΟ λοιπόν, που ε, ασχολείται με την καταστολή των επαναστατικών δυνάμεων, εμείς ασχολούμαστε με μια μεταρρύθμιση μέσω κατάρτισης και εποπτείας. Βασιζόμαστε σε συνεργασία της UPOL με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις αστυνομικές αρχές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ε, γι' αυτό αυτό που μετράει είναι να δούμε την επίπτωση, τη μακροχρόνια επίπτωση της UPOL. Όπως έχω πει στους Αμερικανούς φίλους, βασιζόμαστε στην ε, πραγματογνωμοσύνη και την πείρα μας, την πολυετή μας πείρα στον ε, τομέα της συνεργασίας των αστυνομικών αρχών. Θα έχουμε 300 στελέχη που έχουν 20 τι πείρα. Δηλαδή, ε, μιλάμε ε, για έναν πολύ ψηλό πολλαπλασιαστικό παράγοντα εμπειρίας. Θα πρέπει να μιλήσω και για την ε, αγαστή συνεργασία που είχαμε μέχρι τούδε και μπορώ να σας πω ότι η συνεργασία μεταξύ UPOL, ΕΠΑ και ΝΑΤΟ έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η UPOL και οι δυνάμεις ΝΑΤΟ έχουν προβάλλει μια συνεργασία σε επίπεδο στρατηγίων. Βεβαίως ε, δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση επάνδρωσης καταβάλουμε προσπάθειες να επανδρώσουμε τα, την ε, δομή αυτή με 400, ε, με 400 και πιστεύω ότι θα έχουμε 410 τις επόμενες εβδομάδες που είναι το 70% της ε, προγραμματισμένης επάνδρωσης. Βεβαίω αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά δεν είμαστε και η μοναδική αποστολή στο Αφγανιστάν που αντιμετωπίζει προβλήματα να φτάσει στους ε, απότερους στόχους. Άρα το 75% επάνδρωσης δεν είναι και πολύ κακό. Καταβάλουμε όμως συνεχώς προσπάθειες. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή είναι οι επιμελητιακές δεσμεύσεις που είναι σημαντικές, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να κινηθούμε προς τις επαρχίες. Δεν υπάρχει ευελιξία και υπάρχουν πολλοί όροι για να μπορέσουμε να δράσουμε εκτός Καμπούλ. Αυτό ε, οπωσδήποτε στενεύει τα περιθώρια δραστηριότητας της UPOL, ιδιαίτερα στις επαρχίες. Με βάση, τη διάσκεψη του Λονδίνου, της, με βάση την επικείμενη διάσκεψη του Λονδίνου και επειδή θα υπάρξει και μια μεταβατική περίοδος, δηλαδή μια μετάβαση αρμοδιοτήτων προς τους Αφγανούς, η UPOL θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Και είμαι πεπισμένος ότι με την υποστήριξη των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπάρξει μια εποπτεία της μεταρρύθμισης των αστυνομικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ζητήσω τη βοήθειά σας έτσι ώστε να πείσετε τους συναδέλφους σας στα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και τις κυβερνήσεις των κρατών που εκπροσωπείτε να μας βοηθήσετε στην επάνδρωση αυτή. Αυτό είναι ζωτικής ε, σημασίας ε, γιατί ε, είναι, έχει μεγάλη σημασία για την αξιοπιστία μας και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας πλήρως. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου. Inviting me to... σας ευχαριστώ που με καλέσατε στη συνάντηση αυτή. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω τι συμβαίνει, τουλάχιστον μέσα από τη δική μου οπτική γωνία στο Αφγανιστάν. Ξεκίνησα ε, στην αποστολή αυτή πριν από 15-16 μήνες, όταν η Γιούπολ ακόμα δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα σεβαστή. Υπήρχαν πολλά ιστορικά προβλήματα βασικά από πλευράς επιμελητίας. Και αυτό που χρειάστηκε να κάνω είναι να αποδείξω ότι είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε, είμαστε σε θέση να αποτύχουμε αποτελέσματα. Ένα από τα πρώτα λοιπόν στοιχεία ήταν ότι εξετάσαμε με τους ε, συνεργάτες μας, με τους εταίρους μας ένα πρόγραμμα Δημοτικής Αστυνομίας το Δεκέμβριο του 2008. Εξετάσαμε την πόλη του Ισκαμπούλ για να δούμε τι μπορούσε να γίνει από πλευρά επικοινωνιών, ασφάλειας και ένα από τα στοιχεία ήταν να δημιουργηθεί μία ασπίδα με συντονισμένα σημεία, σημεία ελέγχου μεταξύ της Καμπούλ και των, ε, του εσωτερικού της. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Επίσης, δημιουργήσαμε κινητά μία ελέγχου, επιθεώρηση των σημείων ελέγχου και εκπαιδεύσαμε, πάρα πολλούς ε, νέους ε, αστυνομικούς για τον έλεγχο των σημείων ελέγχου και για τον εντοπισμό ενδεχόμενων ε, καμικάζι. Και είναι πολύ συγκεκριμένο το προφίλ τους. Συγκεκριμένη ηλικία τους, συγκεκριμένη εμφάνισή τους. Και με τον τρόπο αυτό ήταν πολύ πιο επιλεκτικές ε, η επιλεκτική έλεγχη που κάναμε. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί φυσικά θα πρέπει να συνεχίσει και η κυκλοφορία σε μια πόλη όπως η Καμπούλ. Ήταν τεράστια η επιτυχία αυτή και το λέω αυτό επειδή και εμείς ε, ιδρύσαμε το σύστημα αυτό, αλλά και επειδή πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν έρθει στην Καμπούλ και πριν από 6 έως 8 μήνες, αλλά και τώρα μπορούν να δουν σαφώς τη διαφορά. Και μία από τις επιτυχίες μας ήταν όταν έγιναν προεδρικές εκλογές και μιλώ πάντα για επιτυχία σε ό,τι αφορά την αστυνομική συμπεριφορά, έτσι. Δεν μιλάω για γενικότερη επιτυχία. Υπήρχαν λοιπόν δύο-τρει βομβιστέ αυτοκτονία, δύο-τρεις ε, καμικάζοι έτοιμοι να δράσουν και η αστυνομία κατάφερε είτε να του συλλάβει είτε να του ε, σκοτώσει πριν ε, προχωρήσουν στις επιθέσεις αυτοκτονίας. Και τώρα αυτό το σύστημα εφαρμόζεται σε άλλες πόλεις, στο Αφγανιστάν, στο Ιράτ, στην Καταχάρ. Μας έχει δώσει σχετικέ εντολέ στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να καταδείξουμε και στους ετέρους μας, αλλά και σε άλλες χώρες και στα κράτη-μέλη ότι είμαστε σε θέση να πετύχουμε αποτελέσματα. Δεν ήταν μόνο γραφειοκρατία. Κάτι πετύχαμε. Πέραν αυτών, εξετάσαμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Επειδή το ένα τμήμα της αποστολής μας είναι το κράτος δικαίου, αλλά έχουμε τρεις στόχους και το πιο σημαντικό είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Και στο σημείο αυτό η UPOL μαζί με τη συστικά με την UNDP και τους καθεξής ε, ενίσχυσε ένα τέτοιο πρόγραμμα σε όλο το Αφγανιστάν. Για να πω τι συμβαίνει τώρα. Τώρα βρισκόμαστε σε μία φάση συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου εσωτερικών για θέματα συνεργασίας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και υπάρχουν ε, πολλές περιπτώσεις που εξετάζονται ε, από τη UPOL και από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι υποθέσεις αυτές αφορούν και υπουργούς, για παράδειγμα. Και πρέπει αφετέρου να καταδείξουμε στο κοινό ότι καταπολεμούμε και την διαφθορά. Και ξεκινήσαμε λοιπόν μια ενημερωτική εκστρατεία στον τύπο και με μεγάλες αφήσει στην Καμπούλ που αναφέρει έναν αριθμό που μπορούν να καλέσουν οι πολίτες το 199 για την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης έχουμε συσκευές ε, παρακολούθησης, πολύ προηγμένες. Έχουν ήδη γίνει 26 συλλήψεις. Φυσικά οι συλλήψεις αυτές είναι πάρα πολύ λίγες, αλλά ξέρουν πλέον όσοι τροδοκούνται ότι υπάρχει κάποιος που τους παρακολουθεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εκστρατεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς ο αριθμός 199 και θα προωθήσουμε και τις ε, φήμες αυτές για να ξέρουν δηλαδή οι υπέτοι ότι μπορεί και να συλληφθούν, μπορεί και να τους ε, καταδώσουν. Όλα αυτά χάρη στη συνεργασία όλων των εταίρων. Δεύτερος στόχος, η συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και εισαγγελέων. Είναι καινούργιο το σύστημα αυτό. Ένα σύστημα το οποίο πολύ σιγά σιγά έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου στο Αφγανιστάν όπως θα έπρεπε. Είναι μεγάλη λοιπόν. Είναι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό όμως. Και προγραμματίζουμε σχετική συνεργασία και με το Φιλανδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων για την εκπαίδευση αστυνομίας σε ό,τι αφορά θέματα συνεργασίας προκειμένου τα αποδεκτικά στοιχεία να μεταφέρονται δεόντως τους εισαγγελείς και προκειμένου και οι εισαγγελείς να ξέρουν πώς μπορούν να συνδράμουν στο έργο των αστυνομικών. Το τρίτο αφορά, ο στόχος αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών. Σήμερα από τους 96.000 αστυνομικούς μόνο οι 500 είναι γυναίκες. Και αυτό γιατί δέχονται πιέσεις και απειλές επειδή είναι αστυνομικοί και επειδή είναι γυναίκες αστυνομικοί. Είναι δηλαδή πολύ πιο επικίνδυνο να είναι κανείς να είναι κάποια γυναίκα αστυνομικός. Πολλές γυναίκες αστυνομικοί έχουν εκτελεστεί από τα Λιμπάν. Εμείς από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε λάβει εντολή να εφαρμόσουμε σε όλο το Αφγανιστάν μία δομή αντίστοιχη και δίκαιη για τα δύο φύλλα και να δημιουργήσουμε και ένα σύστημα υποβολής αναφορών προκειμένου σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να υπάρχουν σχετικές αναφορές. Φυσικά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πρόθυμο να δεχτεί πιο πολλές γυναίκες για να αυξηθεί ο αριθμός τους μέχρι το 2014 σε 5.000. Είναι πραγματικά τεράστιο το έργο αυτό και φυσικά εξετάζουμε τρόπους για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχουν και γυναίκες αστυνομικοί στα αστυνομικά τμήματα, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες δεν αναφέρουν εγκλήματα σε άντρες θέλουν να μιλήσουν σε μια γυναίκα. Αλλά όπως σας είπα και σε αυτόν τον κλάμπ δραστηριοποιούμαστε με καλή συνεργασία με τις ίπα και με άλλες χώρες μέσω διμερών προγραμμάτων. Από αστυνομικής πλευράς θα πρέπει να βελτιώσουμε να βελτιώσουμε τις ικανότητες των ε, των αντιμετώπισης εγκλήματος. Τεράστιο και αυτό το έργο. Έχουμε τους, ε, τους ε, αστυνομικούς με κάποια ειδίκευση, αλλά όχι με ιδιαίτερη εκπαίδευση. Και αν δείτε στην τηλεόραση, στον τύπο, ε, εικόνες από επιθέσεις αυτοκτονίας, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η σύγχυση, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Βλέπουμε του αστυνομικού να περιφέρονται χωρί να ακολουθούν του κανόνε για την ε, συλλογή αποδεκτικών στοιχείων και μα έχει δώσει εντολή το Υπουργείο Εσωτερικών να εκπαιδεύσουμε την αστυνομική μονάδα καταπολέμηση του εγκλήματο, να κάνουμε εκ νέου εκπαίδευση, να αλλάξουμε τη δομή του τμήματος. Είναι τεράστιο το έργο αυτό που έχει αναλάβει η EUPOL. Πάντα σε συνεργασία με τους εταίρους μας με τις άλλες αποστολές. Κατά δεύτερον, οι μυστικές υπηρεσίες. Κοιτώντας το σύστημα μυστικών υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, εντό τη της αστυνομίας υπάρχουν τέσσερα συστήματα μυστικών υπηρεσιών που δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες κατά της τρομοκρατίας, κατά των ναρκωτικών, των ναρκωτικών και άλλες δύο μονάδες, οι οποίες λειτουργούν όλες αυτόνομα. Και η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται σε θελούσια βάση, όχι σε προχωρητική βάση. Και επίσης έχουμε και το εθνικό, την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και τους, το Σύστημα Βυστικών Υπηρεσιών του Αφγανικού Στρατού πριν από κάποιους μήνες προσπάθησα να συγκαλέσω μία συνάντηση των εταίρων αυτών για να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Ναι, μου ζήτησαν να εξηγήσω τις δημογραφίες που χρησιμοποιώ. Η σύστακα είναι η αμερικανική αποστολή που ασχολείται με την εκπαίδευση του Αφγανικού στρατού και της Αφγανικής αστυνομίας. Η σύστακα λοιπόν είναι Αμερικανική αποστολή, το ίδιο και η ΑΜΚΟ. Τώρα, κάνουμε και συλλογή πληροφοριών και μία υπηρεσία συλλογής πληροφοριών και η μονάδα αυτή συντονίζεται με όλες τις υπόλοιπες. Έχει μόλις γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, πρόταση διότι κατάλαβαν ότι μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Έπειτα έχουμε ένα άλλο σύστημα που στοχεύει σε στενότερη συνεργασία μεταξύ των συλλεκτών πληροφοριών και των αστυνομικών. Πριν γίνει κάτι, όχι μετά. Το σύστημα αυτό ελπίζουμε να εφαρμοστεί στο επόμενο πρόγραμμα, δηλαδή μετά την εφαρμογή της εκπαίδευσης που θα κρατάει δύο μήνες, ώστε να μαθαίνουν ε, και του άλλου μαθήματος που θα αποφεύγει τις δολοφονίες αστυνομικών. Γιατί όλοι όσοι θα συλλέγουν τις πληροφορίες και θα τις επεξεργάζονται μετά, πρέπει να καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα πολύ ψηλότερης ποιότητας από αυτό που έχουμε τώρα. Με τη συνεργασία όλων των προγραμμάτων που σας ανέφερα, των πεζοναυτών, του Σύστακα και άλλων. Έχουμε και τη μονάδα του ελέγχου και ανταπολέμησης της εγκληματικότητας που το λέμε PCCC ή P3C. Γιατί έτσι θεωρούμε ότι όταν κάποιος παίρνει μια διαταγή δεν ξέρει και πώς να την εφαρμόσει και οι περισσότεροι δέχονται εντολές από το Υπουργείο Εσωτερικών οι αστυνομικοί. Όλα πρέπει να τα εγκρίνει πρώτα το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό δεν είναι σωστός τρόπος λειτουργίας της αστυνομίας. Πρέπει η αστυνομία να έχει όλους τους πόρους που διαθέτει για να λύσει το πρόβλημα χωρίς να απαιτούνται ανδιάμεσες εγκρίσεις. Και έτσι έχουμε τους τέσσερις πυλώνες της αφγανικής αστυνομίας που σας ανέφερα. Του ελέγχου στα σύνορα, του αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, των ναρκωτικών κλπ. Προβλέπετε και ένας πέμπτος πυλώνας, ακόμη δεν έχει όμως συζητηθεί και δεν θα σας τον αναφέρω. Σας είχα ήδη πει προηγουμένως ότι είχε υπάρξει και το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε με αφορμή τις εκλογές όπου 20.000 άνθρωποι είχαν πάρει μαθήματα ως προς τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς μιας δημοκρατικής αστυνομίας στα εκλογικά τμήματα. Και μετά κάναμε και μια αξιολόγηση. Φέρθηκαν όπως έπρεπε έλεγξε και ο υπεύθυνο στρατηγός Μορλάν της ε, αποστολής της Ένωσης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αστυνομία είχε αποτελέσματα από καλά μέχρι εξαιρετικά καλά στην Καμπούλ και στο κέντρο. Ανατολικά υπήρξαν μερικά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι καθήκον μας να πούμε στην Αφγανική αστυνομία ότι όσο και να σας επικρίνουμε εκείνη την ημέρα φερθήκατε πολύ καλά. Και την περασμένη Δευτέρα που έγινε η επίθεση στην Καμπούλ, η A&A και η A&P αντιμετώπισαν το πρόβλημα. Μόνοι τους. Και πολύ καλά. Δεν ξέρω αν μήπως εξαντλήθηκε ο χρόνος μου, μήπως. Α, όχι λοιπόν. Και τώρα θα ήθελα η αποστολή αυτή να εφαρμόζεται σε όλο το Αφγανιστάν και όχι μόνο στην Καμπούλ. Να καλύπτει το σύνολο της επικρατείας. Αλλά γι' αυτό χρειάζομαι και τη βοήθειά σας διότι έξω από την Καμπούλ, πέρα από την Καμπούλ, χρειαζόμαστε στέγαση των λεγόμενων PRTs και χρειαζόμαστε και την ασφάλειά τους των PRTs και το προσωπικό των PRTs και ελαστικότητα για, από τα κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη χορηγούν ορισμένους αξιωματικούς ή αξιωματούχους στην Καμπούλ και στη γύρω περιοχή, αλλά σε άλλα PRTs δεν έχουμε στέγαση. Τι να κάνουμε να κατασκηνώσουμε. Υπάρχουν τρεις-τέσσερις χώρες που μας δίνουν και τη στέγαση, αλλά οι υπόλοιπε για πολιτικούς μάλλον λόγους δεν επιδεικνύουν τέτοια ελαστικότητα, ενώ είναι απαραίτητη. ενώ χρειαζόμαστε κόσμο και έξω από την Καμπούλ. Αλλιώς θα πρέπει να πούμε στην CPCC ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά που μας ε, παραγγείλατε. Γιατί η Γιούπολ ορισμένα μέλη θεωρούν ότι πρέπει να σταματήσει ενώ έχει δείξει ότι φέρνει αποτελέσματα και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα συνεχίσει να φέρει αποτελέσματα αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ παραπάνω από όσα μέσα διαθέτουμε που δεν μας τα χορηγείται. Αν υπάρξει αυτή η ελαστικότητα που σας είπα και η στέγαση και το προσωπικό τότε θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους μας σε ολόκληρο το Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας γιατί παραβρίσκεστε εδώ και για να σας τιμήσω διότι η UPOL τα κατάφερε πολύ καλά σε σχέση με διάφορες άλλες διεθνείς αποστολές στο Αφγανιστάν που δέχονται επικρίσεις. Εσείς σταθήκατε επαγγελματίες, κύριε Βιτρούπο, δεν μπορούμε παρά να σας συγχαρούμε, γιατί κάτω από δύσκολες συνθήκες ανταποκριθήκατε στην αποστολή αυτή της UPOL. Πριν γίνει ένας γύρος του τραπεζιού, θα ήθελα να σας ρωτήσω με μια μεσότητα ορισμένα πράγματα, διότι πιστεύω ότι υπάρχει μία απογοήτευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι πολλοί εμπλεκόμενοι διεθνείς φορείς έχουν παρευρεθεί στο Αφγανιστάν. Ε, σε εμά βλέπουμε ότι υπάρχει μία διάχυση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, είτε μονομερός, είτε σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και ούτω καθεξής υπάρχει μια απογοήτευση σε σχέση με την ε, περιορισμένη εμβέλεια της UPOL ποσοτικά σε σχέση με τις διεθνείς προσπάθειες και σε σχέση με αυτή την πληθώρα παρεμβάσεων διεθνών φορέων, γιατί κύριε Βίτρουπ συνεργάζεστε κι εσείς μαζί τους και επειδή πρόκειται για ένα περίπλοκο ε, νήμα φορέων στο Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστείτε με διάφορες διευθύνσεις της αστυνομίας στο Αφγανιστάν. Ε, έχουμε λοιπόν την τάση να σας ρωτήσουμε μία αποστολή τόσο περιορισμένη ποσοτικά μπορεί να δράσει. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της UPOL σε σχέση με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ ή τις αποστολές των ΙΠΑ ιδιωτικές ή δημόσιες που προβαίνουν στην κατάρτιση των τοπικών φορέων. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της αποστολής Πολ. Αυτή είναι μια άμεση, ε, μια ερώτηση με μια κάποια αμεσότητα. Ο... Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέρμαν και μετά στους διάφορους συντονιστές θα πρέπει να είσαστε αρκετά συνεκτικός για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Merci beaucoup, monsieur. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Έτσι ώστε ο κύριος Βίτρουπ να βγάλει τα ακουστικά του. In English, uh, for you, uh, Θα τα πω στα αγγλικά. Συμφωνώ και επαυξάνω το θαυμασμό για αυτά που κάνατε, γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρατε να δώσετε στη Γιούπολ την ε, ισχύ, την ε, δομή που έλειπε στην αρχή. Όλοι συμφωνούμε από αυτού και ήταν πραγματικά δύσκολο το έργο σας. Και νομίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ευρεία συνένεση για την ανάγκη υποστήριξης της αποστολής σας. Ωστόσο, θα ήθελα να μας απαντήσετε στην ε, πρώτη ερώτηση του Προέδρου σε ό,τι αφορά δηλαδή την προστιθέμενη αξία της UPOL, σε ό,τι αφορά τις εργασίες και τις εκπαιδεύσεις του ΝΑΤΟ και των ε, ΙΠΑ. Εξετάζοντας λοιπόν την κατάσταση σήμερα στο Αφγανιστάν και στη Σύνοδο του Λονδίνου θα γίνει ανάλογη ανάλυση, βλέπουμε φυσικά ότι υπάρχουν αρνητικά και θετικά στοιχεία. Θετικά στοιχεία η εκπαίδευση, 6 εκατομμύρια παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, ένα τρίτο είναι κορίτσια, το υγειονομικό σύστημα, οι υποδομές, δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί και ούτω καθεξής. Στην αρνητική, αρνητικές, τα αρνητικά στοιχεία είναι πιο πολλά, πολύ φοβάμαι. Πολύ πιο πολλά. Αυξάνονται τα περιστατικά βίας και τα στρατεύματα δεν επηρεάζουν την κατάσταση αυτή. Η Αλκάιντα, η Ταλιμπάν και το κόστος ε, των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι σήμερα 200 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ε, δολάρια το έτος. Και των οποίων ε, μεγάλο μέρος καλύπτονται από τις ΗΠΑ. 200 δισεκατομμύρια δολάρια λοιπόν για ένα σύστημα ασφάλειας το οποίο αποτυγχάνει τελικά, το οποίο έχει επανέλθει. Η διαφθορά αφορά τους μισούς Αυγανούς σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του UNODC πολλοί πολίτες πέφτουν θύματα των ενεργειών αυτών και αυτό κλονίζει την εμπιστοσύνη σε μας στη Δύση. Κλονίζεται λοιπόν και η εμπιστοσύνη και στη δική μας συμμαχία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και δεν είναι τυχαίο ότι το διοργανώνεται η στο Λονδίνο. Και είναι κρίμα που η κυβέρνηση η Βρετανική δεν κάλεσε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά το γεγονός ότι διδραματίζουμε ένα σημαντικό, αν και μικρό, ρόλο. Είναι λοιπόν κρίμα που δεν θα συμμετάσχουμε και μου προκαλεί και έκπληξη. Αυτή η διάβρωση όμως της εμπιστοσύνης του τι κάνουμε στο Αφγανιστάν θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε πιο πολύ εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική της Αμερικανικής κυβέρνησης που θέλει λιγότερη στρατιωτική παρέμβαση και πιο πολύ πολιτική παρέμβαση. Και νομίζω ότι είναι λάθος να πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να εφαρμόσουμε στο Αφγανιστάν τις ίδιες λύσεις όπως ε, στο Ιράκ. Γιατί αν ε, ρωτήσουμε τον στρατηγό θα μας πει ότι πρέπει να στείλουμε πιο πολλούς στρατιώτες. Γιατί αυτός ε, είναι ο κλάδος τους. Δεν έχω χρόνο να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Αυτό που είναι σημαντικό ωστόσο είναι να επενδύσουμε στο Αφγανιστάν. Την ασφάλεια δεν θα την πετύχει μόνο η αστυνομία και ε, ο στρατός και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομική ανάπτυξη, στην γεωργία, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, όπως πολύ σωστά ορίζει τους στόχους αυτούς η νέα αμερικανική πολιτική. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Αυτό σημαίνει επίσης πιο πολλές μικροπιστώσεις για τους Αφγανούς που θέλουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και τις φιλοδοξίες τους. Σημαίνει καταπολέμηση της διαφθοράς και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η Γιούπολ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την Γιούπολ, γιατί αυτή η πολιτική προσέγγιση δεν θα λειτουργήσει ποτέ χωρίς μια ναι. ισχυρή αφγανική αστυνομία, αλλά θα πρέπει να δοθεί και ένα τέλος στην ε, ατιμορρησία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στο Αφγανιστάν, που ναι μεν υφίστανται, αλλά δεν έχουν ακόμα ιδιαίτερη ισχύ. Να ενισχύσουμε τις τοπικές ε, κυβερνήσεις, να ενισχύσουμε τους θεσμούς. Και είναι θετικό που αποφασίστηκε να αναβληθούν οι εκλογές για την 18η Σεπτεμβρίου. Γιατί αρχικά προβλέπονταν για τις 22 Μαΐου. Αυτό είναι καλό νέο γιατί θα μπορέσουν έτσι να γίνουν κάποιες απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρξει μία ανεξάρτητη επιτροπή εκλογική. Να υπάρχει και ένα μητρό του εκλογικού σώματος και φυσικά να αποκλειστούν οι υποψήφοι με ποινικό μητρό από το Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν πριν τις 18 Σεπτεμβρίου. Αν θέλουμε να σταθούμε επιτυχία οι εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα πρέπει να εντάξουμε τις προσπάθειες αυτές που καταβάλλεται για την εκπαίδευση της αφγανικής αστυνομίας. Δεν θα είναι εύκολη ούτε γρήγορη η διαδικασία, η εκπαίδευση αγράμματων αστυνομικών, αλλά θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ασκήσουμε πίεση και στις κυβερνήσεις μας για να υποστηριχθεί και η επάνδρωση της UPOL και το θέμα της ευελιξίας που θίξατε και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουν τώρα οι εκπρόσωποι των ομάδων. από τους τέσσερις εμπειρογνώμονες, μετά τους τέσσερις εμπειρογνώμονες κάθε φορά θα γίνεται ένα γύρος ερωτήσεων και παρακαλώ τις ερωτήσεις να τις θέτετε ανάλογα με το θέμα, όχι ο καθένας για τα πάντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κλόπενχάουερ, είπατε στην αρχή ότι η συνεργασία έχει βελτιωθεί κατά πολύ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Να συμπεράνω, λοιπόν, ότι η μη υπογραφή της τεχνικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και στη συνεργασία επιτόπου. Δεύτερη ερώτηση. Αναφέρθηκε ήδη ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, υπάρχουν επίσης εθνικές αποστολές εκπαίδευσης από τις εθνικές κυβερνήσεις. Πώς ε, διαιρούν και κατανέμουν τις αρμοδιότητες τις αυτές. Ποιοι δηλαδή είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση και ποιοι συντονίζουν τις δράσεις. Έχετε αριθμητικά στοιχεία. Διάβασα κάπου ότι θα προσθεθούν και 169 τοπικές δυνάμεις στις 400 δυνάμεις που υπάρχουν ήδη και πώς θα υπάρχουν, πώς θα συνεργαστούν αυτές οι δυνάμεις ύστερα. Πώς γίνεται η εκπαίδευση από τις εθνικές κυβερνήσεις. Ακούσαμε ότι υπάρχουν ε, στρατιωτικές αστυνομίες, συνοριοφύλακες και ούτω καθεξής. Έχουν πραγματικά την εκπαίδευση που χρειάζονται. Και τελευταίο στοιχείο για τις πληρωμές. Νομίζω ότι ξέρουμε ότι από όλες τις περιοχές που υπάρχουν κρίσεις, ότι δεν εγγυώνται οι πληρωμές. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι συχνά οι αστυνομικοί μπορεί να αλλάξουν πλευρά. Πώς μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε το θέμα αυτό των πληρωμών των αστυνομικών. Grazie συνάδελφος Γκάλερ υπέβαλε ορισμένες από τις ερωτήσεις που θα ήθελα να απευθύνω και εγώ. Συμφωνώ με όσα ανέφεραν οι δύο εισηγητές, διότι στην πραγματικότητα η Ιούπολ, μάλλον η Ιούπολ ε, δέχεται πολλές επικρίσεις άδικες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες ε, αυτής της αποστολής από στρατηγικής πλευράς. Σε σχέση με τη συνεργασία με τις αφγανικές αρχές και αστυνομία. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω εξ ονόματος της ομάδας μου ότι υποστηρίζουμε τη δράση της UPOL. Βεβαίως υπάρχουν και ορισμένα ερωτηματικά, τα οποία υπενθύμησε και ο πρόεδρος Ντανζάν και ο συνάδελφος Γκάλερ. Θα ήθελα να επενθυμίσω ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ως προς την, τις σχέση ασφάλειας που διέπουν τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, που προέβαλε ο συνάδελφος Γκάλερ, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε μία επιμέρους πτυχή, διότι μιλάμε για 245 όχι για 520 συνολικά. Πώς θα φτάσετε στους 310 και εάν φτάσουμε τους στόχους των 400 πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση γιατί μιλάμε και για, ε, πολλά, και για ένα παρεπόμενο μάλλον κόστος. Όπως είπε και ο πρόεδρος Ντάνζαν, αυτό που έχει σημασία είναι και η προστιθέμενη αξία. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο η αξιέπαινη αυτή εργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς μπορεί να προωθηθεί χωρίς να ε, αντιμετωπίσουμε και, το δικαστικό, και τη δικαστική πτυχή. Δηλαδή ένα δικαστικό σύστημα, ένα δικαιοδοτικό σύστημα. Πώς αντιμετωπίζει η UPOL το θέμα μιας ε, γενικότερης δικαιοδοσίας και δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες. Τέλος, ως προς τις ε, χρονικές προοπτικές αυτής της αποστολής, πώς ε, κρίνονται. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, τοπική παράδοση. Επίσης, πώς βλέπετε την παρουσία των ΙΠΑ, όπως είπε και η Υπουργός Εξωτερικών Κλίντον, Περάσαμε από τους 320 στους 1000 Αμερικανούς που παρίστανται στον τομέα πολιτικών υποθέσεων και όχι στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πώς ε, προβλέπετε, ε, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή, τη συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, αυτό το Civil Surge. Ευχαριστούμε. Ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο μιλητές, Κλόπενάουρ και Βιτρούπ, τα εξή. Βοηθούμε τους Αφγανούς. Θα πρέπει να τα καταφέρουν βεβαίως μόνοι τους σε σχέση με τις αστυνομικές αρχές. Άρα, ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια, ένα γενικότερο όραμα της ε, αφγανικής κυβέρνησης και πώς μπορεί να τεθεί στην πράξη, διότι εσείς μιλήσατε για το γεγονός ότι ως προς την αστυνομία και την αστυνομική συνεργασία εμπλέκονται πολλά υπουργεία. Πώς ε, έχει αυτή η συνεργασία, επεκτείνεται σε επαρχίες ή σταματάει στην Καμπούλ. πώς αποτελεσματικές είναι αυτές οι αρχές. Και τέλος, γίνονται ακροάσεις στο Αφγανικό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη δραστηριότητα πολλών υπουργών της κυβέρνησης Καρζάη. Η διοργάνωση της αστυνομίας, η οργάνωση της αστυνομίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των συζητήσεων. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, εκφράσατε την δέσμευση της ε, UPOL και συμφωνώ απόλυτα με την εμπιστοσύνη αυτή που εκφράσατε και να ευχαριστήσω και τους ε, ομιλητές για την ε, πολύ ε, καλή παρουσίαση του έργου τους εκεί, που είναι σημαντικό αλλά και σίγουρα δύσκολο. Αλλά για να μην μείνουμε μόνο στα θετικά. Να πω ότι συμφωνώ και με την κάποια απογοήτευση που εκφράστηκε. σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει ως τώρα μετά από όλες ε, τις ε, προσπάθειες της UPOL. Θεωρώ ότι δεν προχωράμε αν είμαστε απλά ευγενικοί ο ένας με τον άλλον. Ο Τόμ Κιόνιξ, ο πρώην επικεφαλής ε, της, της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, υπέδειξε πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες στον τύπο στη Γερμανία ότι ο αριθμός των αστυνομικών δυνάμεων των 400 δηλαδή αστυνομικών δεν είναι επαρκής. Είπε πολλές φορές ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2.000 τέτοιες δυνάμεις. Το κόμμα, το κόμμα μου πολέμησε και αγωνίστηκε για να αποσταλούν πιο, πολλές, ε, πιο πολλοί Γερμανοί αστυνομικοί. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποσταλθούν πιο πολλοί Γερμανοί στρατιωτικοί στο Αφγανιστάν από ότι είναι συνολικά από όλη την Ευρώπη στο Αφγανιστάν. Δεν δέχομαι λοιπόν να ωρεοποιούμε την ε, κατάσταση και να ξοραίζουμε τα πράγματα. Ο στόχος είναι πολύ πιο υψηλός και είναι πραγματικά ντροπή. Και νομίζω ότι πριν από την σύνοδο του Αφγανιστάν στο Λονδίνο θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να δούμε αν κάνουμε μια θεωρητική πολιτική και δεν θέλω να αμφισβητήσω το έργο των ε, δυνάμεων ε, στο Αφγανιστά αυτό που θέλω να αμφισβητήσω είναι τη δέσμευση της Ευρώπης. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποιες χώρες επιδεικνύουν ε, περιορισμένη ευελιξία. Ποιες χώρες είναι αυτές που δεν αποστέλουν αρκετές αστυνομικές δυνάμεις. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να ασκήσουμε τέτοια πολιτική. Και αυτό που είπε και ο κύριος Γκάλερ δικαίως, τίθεται θέμα πληρωμή των αστυνομικών. Δεν έχει νόημα να του εκπαιδεύουμε και μετά να μην μπορούμε να τους πληρώσουμε και να φεύγουν να δουλέψουν για εμπόρους ναρκωτικών κτλ. Έχει γίνει πρόταση να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πληρωμές των αστυνομικών. Δεν θα ήταν μεγάλο το ποσό. Και τώρα συζητάμε το ενδεχόμενο να αγοράσουμε τους Ταλιμπάν. Δεν συζητήσαμε όμως, δεν καταφέραμε να αποφασίσουμε την χρηματοδότηση των αστυνομικών που εκπαιδεύουμε. Θα ήθελα να έχουμε λίγο πιο υψηλές ε, φιλοδοξίες και σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευόμενους εκεί, γιατί στη τελική ανάλυση η αποστολή αυτή είναι αποστολή Καμπούλ. Και είπατε απολύτω ε, δικαίω ότι δεν θα πρέπει να παραμείνει αυτή η αποστολή, η αποστολή τη Καμπούλ. Θα πρέπει να είναι δίκαια τα πράγματα και θα πρέπει να θέσουμε να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα εξ ονόματο του Κοινοβουλίου. Ja, vielen Dank. Η κυρία Λόζινγκ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναφερθώ σε αμυγός στρατιωτικά ζητήματα γιατί η ανάλυση του ρόλου της αστυνομία σε κάθε τόπο μπορεί να αποτελεί και μία ανάλυση των κοινωνικών συγκρούσεων. Προϋποθέτει, προϋποθέτει και τον ρόλο των αστυνομικών. Να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπέρμαν. Νομίζω ότι υπάρχουν και μελέτες που καταδεικνύουν τη σχέση της ανεργίας της φτώχειας που δημιουργούν και υποθάλπτουν τις επικίνδυνες καταστάσεις εκεί. Δεν θα επεκταθώ όμως στο σημείο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι αυτά τα θέματα αφορούν και την εικόνα της αστυνομίας. Έχω την αίσθηση ότι κάπως ε, ωρεοποιούμε τα πράγματα. Μιλάμε πραγματικά για αστυνομία ποινική ε, δίωξης. Είπατε πώς πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία σε μια δημοκρατία. Μα δεν είναι δημοκρατία. Με ποιο τρόπο συμμετέχει και η αστυνομία σε συγκρούσεις που προέρχονται από πολίτες. Μπορούμε να διαχωρίσουμε το πολιτικό σκέλος από το στρατιωτικό σκέλος. Σας ερωτώ λοιπόν, πόσο συμμετέχει η αστυνομία σε θέματα κατάπνιξης των εξεργέσεων που προκύπτουν για παράδειγμα από τις συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και παστούν. Αυτό είναι στρατιωτικό καθήκον. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες των συγκρούσεων για να ξέρουμε καν ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της αστυνομίας εκεί. Να κάνω όμως και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ρώτησαν πολλοί συνάδελφοι το θέμα του κόστους. Νομίζω ότι και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Κατά το παρελθόν, ο εξοπλισμός ε, τον Ταλιμπάν, για παράδειγμα, χρηματοδοτούνταν και από, την, από τη ΣΥΠΑ. Θα ήταν πραγματικά παράνοια να συνεχίσουμε τέτοιες διαδικασίες, να γίνεται δηλαδή εκπαίδευση από τη UPOL αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες δεν πληρώνονται μετά και μετά να πηγαίνουν στους Ταλιμπάν. Να ρωτήσω λοιπόν, πόσο θεωρείτε ότι είναι το κόστος για τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας και από πού θέλουμε να προέλθει η χρηματοδότηση του κόστου αυτού. Ο κύριος Κλόμπενχάουρ, αν δεν κάνω λάθος, ανέφερε την αλλαγή των ε, στόχων της αστυνομίας. Ποιες αλλαγές είναι αυτές και ποιοι είναι οι στόχοι που θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχει αστυνομία και άλλη μια συγκεκριμένη ερώτηση. για την επέκταση της επάνδρωσης της UPOL. Merci, um, Σε αντίθεση με τον κύριο Μπέρμαν, θα ήθελα να πω ότι δεν ε, κληθήκαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι μάλλον δεν κληθήκαμε και χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία. Το Μάιο του 2008 παρευρέθηκα εγώ εκεί, αλλά οι θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας του ΝΑΤΟ, εδώ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μας επέτρεψαν να δούμε τι δεν πάει σωστά με το Αφγανιστάν. Στο μεταξύ άλλαξαν τα πράγματα, ήρθε ο πρόεδρος Ομάμπα Ομπάμα και έχει αλλάξει αυτή η ορθοδαξία. Και έτσι ακολουθούμε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές που θέλαμε, την ανθρώπινη ασφάλεια, την προστασία του πολίτη, την ε, ανάπτυξη του Αφγανιστάν. Η ερώτησή μου έχει ως εξής. Κατανοώ τη μεγάλη σας προσπάθεια με μεγάλους κινδύνους υπέρ της υποστήριξής σας, αλλά θα πρέπει να συμμετέχετε σε μια ευρύτερη στρατηγική που να είναι απόλυτα λογική. Θεωρείτε ότι η στρατηγική προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει διαφορά, αποτελεί πραγματική διαφορά σε σχέση με την προσέγγιση των ΗΠΑ ως προς την ασφάλεια και την δημιουργία κράτους στο Αφγανιστάν. Δημιουργία κρατικών υποδομών. Τι γίνεται στον ε, δικαιοδοτικό τομέα. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την αστυνομία, μιλάμε για ένα δικαιοδοτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν. Όταν παρευρέθηκα εκεί έμαθα ότι η γενική η οι εισαγγελείς και οι δικαστές πληρώνονταν λιγότερο από τους αστυνομικούς, υπήρχε διαφθορά και είναι ιδιαίτερα διεφθαρμένοι. Στις φυλακές υπάρχουν ε, όχι εγκληματίες αλλά γυναίκες πρωτίστως. Και εσείς μας είπατε ότι υπάρχουν 500 μόνο γυναίκες στις ε, αστυνομικές αρχές στο Αφγανιστάν θα πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες ως προς την εξισορρόπηση της παρουσίας των δύο φύλων στην αστυνομία. Ελέγχθη ότι ορισμένες ε, χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να προωθήσουν ε, μία παράπλευρη βοήθεια στη u έτσι ώστε να σας δοθεί ένα input. Όταν βρέθηκα στο Αφγανιστάν, έμαθα ότι υπήρχε μεγάλο χάσμα. Ε, ως προς την ε, μια πραγματική δύναμη, αστυνομική δύναμη και σε σχέση με την προσέγγιση των ΙΠΑ ως προς τη συγκρότηση αστυνομικών δυνάμεων. Η Eurogen 4 θα μπορούσε ίσως να σας βοηθήσει. Πιστεύετε ότι θα συνεισέφερε πραγματικά όταν μιλάτε για το έγκλημα και για την αντιμετώπιση του. πρέπει να δούμε ουσιώδη ζητήματα. Υπάρχει ένα όραμα της αγωνικής κυβέρνησης το οποίο θα πρέπει να συντράβουμε και εμείς. Αυτό είναι μια πραγματική δοκιμή, διότι όταν παρευρεθήκαμε εκεί ρωτήσα τι γίνεται με τη δραστηριότητα του αδελφού του Πρόεδρου Καρζάη, ο οποίος είναι ένας βαρόνος των ναρκωτικών. Έχει φυλακιστεί. Υπάρχουν ε, ουσιώδη ερωτήματα ως προς την αντιμετώπιση του εγκλήματος και την καταπολέμηση των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Ο κύριος ε, Ζέμκε. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίτρου. Ευχαριστώ. Άκουσα τις πληροφορίες αυτές με πολύ μεγάλη προσοχή, διότι πολλά χρόνια ήμουν υπεύθυνο για πολλούς Πολωνούς στρατιώτας που είχαν συμμετάσχει σε αποστολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αλλά προτιμώ να βρίσκομαι εδώ παρά στην Καμπούλ και αλλού. Έχω όμως και τρία ερωτήματα μετά τις παρατηρήσεις αυτές. Καλά μου φαίνονται όλα όσα κάνετε εκεί, ε, αντιμετωπίζετε και πολλούς κινδύνους, αλλά πρέπει να δούμε μήπως υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης. Πρώτον, συμφωνώ και στρατηγέ μου ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι η σύραξη, η διαμάχη διαρκεί πάρα πολύ και δεν έχει επιτευχθεί συντονισμό των, διαφόρων, των προσπαθειών των διαφόρων υπηρεσιών πληροφοριών και πληροφόρησης. Υπάρχουν διάφορες στρατιωτικές υπηρεσίες και αστυνομικές που διαθέτουν πληροφορίες αλλά δεν τις συντονίζουν και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία λογική ανάλυση και δεν χρησιμοποιούνται. Πρώτο λοιπόν ερώτημα, πώς λύνεται το πρόβλημα των μεταφράσεων ας πούμε. Διότι ακούγονται ηλεκτρονικά πολλές πληροφορίες αλλά πρέπει μετά να τις επεξεργαστούν ειδικοί και γλωσσομαθείς που να γνωρίζουν τις τοπικές γλώσσες και διαλέκτους. Γι' αυτό το πρόβλημα το έχετε προσέξει. Δεύτερο ερώτημα. Συμμερίζομαι την άποψη των συναδέλφων που μίλησαν προηγουμένως και εγώ είχα αυτή την εντύπωση στο Αφγανιστάν αλλά και στο Ιράκ ότι, ότι λέγω μερικές χώρες συμπεριφέρονται υπεύθυνα ως προς τη διεθνή ασφάλεια, άλλες όμως, και το λέω με τα συγχωρήσεως, προσποιούνται ότι το πράττουν. Ποιούνται. Δηλαδή δρούν μόνο μέσα στις στρατιωτικές τους βάσεις και ποτέ απ' έξω. Πρέπει λοιπόν νομίζω να επικρίνουμε, να καταργήσουμε αυτές τις ε, ψευτοδραστηριότητες. Τρίτον και σημαντικότερον, η λογική των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν πρέπει να είναι οι εξής δύο τελείες. Τον κυριότερο ρόλο να τον παίζει η αστυνομία, στη βάση της υπόθεσης ότι με τον χρόνο θα καταλήξουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο να μεταβιβάσουν τη, όλες τους τις δικαιοδοσίες στην αστυνομία. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι έχουν υπάρξει, ότι έχουν επιμορφωθεί, εκπαιδευτεί κατάλληλοι Αφγανοί ε, αστυνομικοί διότι στο Ιράκ είδα ότι το 30% των εκπαιδευομένων εγκατέλειπαν τα μαθήματα. Ευχαριστούμε. Ήθελε να προσθέσει κάτι ο κύριος Μπέρμαν τώρα. Θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά που είπε η Άννα Γκόμες. Κατά πόσο ε, δεν ε, είχε ε, νόημα η όλη αυτή η προσπάθεια. κατά πόσο ήταν πραγματικά irrelevant. Βλέπουμε ότι στο Αφγανιστάν φτάσαμε σε μία εισβολή νεοαπικιακού τύπου και αυτή η κληρονομιά των ετών Bush, της κυβέρνησης Bush, θα πρέπει να αλλάξει και να μεταστραφεί σε μία αναπτυξιακή βοήθεια. Βεβαίως χρειάζεται η συνεργασία των αστυνομικών αρχών και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Το 95% των διαφορών επιλύονται σε επίπεδο καλυμπάν, διότι είναι η μόνη που δεν είναι διεφθαρμένη. Είναι η μόνη ε, δικαστική αρχή που δεν είναι διεφθαρμένη. Δηλαδή οι Αφγανοί θα θέλαν να πιστέψουν σε αυτό το σύστημα, αλλά έμπρακτα δεν τους επιτρέπει η διαφθορά. Αυτό θα πρέπει να αλλάξουν οι Αφγανοί με τη δική μας βοήθεια. Ο Καρζάη είναι υπεύθυνος για τις υποσχέσεις που έχει δώσει όταν ανακηρύχθηκε πρόεδρος. Και θα πρέπει να θέσουμε όρους χορήγησης βοήθειας. Δηλαδή, αν δεν επιτεθούμε και δεν καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και την απάτη, τότε καμία βοήθεια δεν θα χορηγηθεί. Ο κύριος Πούσικοφερ. Μία μικρή ερώτηση προς τον κύριο Κλόμπενχάουρ, γιατί ο κύριος Μπέρμαν είπε μόλις ότι προκλήθηκε μία νέα αποκεντρωτική ε, προσέγγιση Θέλω να σας ρωτήσω, η εντολή του ΟΗΕ νομιμοποιείται και στην ε, εντολή της Ευρώπης για τη Γιούπολ. Πού βρίσκεται αυτό το νέο αποκαιοκρατικό αυτό στοιχείο, κύριε Κλόπενάουερ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα αρχίσω εγώ και θα αφήσω στο συνάδελφο την τελευταία πινελιά. Θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Αυτό τουλάχιστον διαισθάνομαι από την Ομίγυρη. Συμμερίζομαι την ανυπομονησία σας. Ε, δεν θα ήθελα να μιλήσω για απογοήτευση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας τέτοια πολυτέλεια. Συνεργαζόμαστε σκληρά με τα κράτη-μέλη για να τύχουμε υποστήριξη στο φθινόπωρο. Καταρτήσαμε λεπτομεριακά σχέδια και με βάση αυτά είμαστε πεπισμένοι ότι θα φτάσουμε στους 310-311 σε σχέση δηλαδή με τους 245 που είχατε στα χαρτιά σας. Δηλαδή θα έχουμε 310, 310 άτομα προσωπικό και έχουμε και το τοπικό προσωπικό, μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης καταβάλαμε προσπάθειες έτσι ώστε η δική μας ε, αστυνομική να πληρώνονται καλύτερα, διότι ε, δυστυχώς δεν υπήρχε καθόλου καλή ε, πληρωμή και ημερήσια αποζημίωση. Έχουμε αυξήσει την ημερήσια αποζημίωση και το έχουμε αυξήσει πάνω από το προσδοκόμενο όριο. Οι αστυνομικοί θα πρέπει να βρεθούν εκεί σε θελούσια βάση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τους υποστηρίξουν. Βεβαίως Υπάρχει ανταγωνισμός και με διμερεί σχέδια ή προγράμματα ως προς την UPOL. Λοιπόν, για να δούμε την ευρύτερη εικόνα. Ως προς την αρχική ερώτηση του Προέδρου, την ύπαρξη προστιθέμενης αξίας. Αυτή η σκέψη μας διακατέχει συνέχεια. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, πόσα χρήματα δαπανώνται, όλα αυτά γίνονται για κάποιο στόχο. Άρα υπάρχει προστιθέμενη αξία. Μπορώ να πω ότι αν δούμε τη νέα αμερικανική στρατηγική που εστιάζει την προσοχή στις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις και αυτός είναι απαράβατος όρος για να επιτύχουμε, νομίζω ότι βρισκόμαστε ε, στην την κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο χώρο. Η πρωταρχική μας αποστολή είναι να βοηθήσουμε την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και να της ε, χορηγήσουμε ένα μέσο πολιτικής ασφάλειας έτσι ώστε να υπάρχει όλα αυτά να εντάσσονται σε μία βιώσιμη στρατηγική επιβίωσης. Εκεί καταβάλουμε προσπάθειες. Άρα δεν, δεν αντιτασσόμαστε σε, στις στρατιωτικές προσπάθειες, απλώς τις ε, συμπληρώνουμε με ένα ζωτικό στοιχείο πολιτικής συνεργασίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάτι άλλο, το χρονικό μας ορίζοντα. Για να επιτύχουμε στην αποστολή μας θα πρέπει να την εντάξουμε χρονικά σε έναν πενταετή και ίσως δεκαετή ορίζοντα, διότι μιλάμε για μια χώρα με πολύ χαμηλό αναπτυξιακό ρυθμό που έχει καταστραφεί μετά από ένα τριακονταετή ε, πόλεμο. Άρα οι περισσότεροι αστυνομικοί είναι αναλφάβητοι. Είναι πολύ δύσκολο να στήσουμε μια λειτουργική αστυνομική δύναμη. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Από το 2007 βρισκόμαστε in situ, άρα η UPOL έφτασε πολύ αργά σε σχέση με την διεθνή επέμβαση μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Άρα εντασσόμαστε κι εμείς, αλλά δεν θα είμαστε έτοιμοι το 2011. Αυτό είναι αδύνατο. Τα καλά νέα είναι, έγινε στο γεγονός ότι παρόλο που μας στοιχίζει αποστολή 64 εκατομμύρια ετησίως, είναι λιγότερο δαπανήρια από μια στρατιωτική επιχείρηση, διότι δεν έχουμε ε, ε, ακριβά, δεν χρησιμοποιούμε ακριβά μέσα και δεν υπάρχει κόστος σε ανθρώπινη ζωή. Άρα αν τα κράτη-μέλη μπορούν να μας υποστηρίξουν, τότε θα έχουμε μία βιώσιμη θα έχουμε να κάνουμε μια βιώσιμη επιχείρηση που θα αντέξει στο χρόνο. Γιατί εκεί πρέπει να εντάξουμε την αποστολή μας. Έτσι πρέπει να την εντάξουμε. Και έτσι θα προσμετρήσουμε και την προστιθέμενη αξία. η αφγανική κυβέρνηση. Γιατί πολλές φορές πρέπει να πείσουμε τους ομόλογους να κάνουν κάτι έμπρακτα. Άρα ε, επιβραδύνεται η όλη στρατηγική. Και πολλές φορές ε, δεν γίνεται κατανοητό αυτό εύκολα, διότι χρειάζεται χρόνο. Um, Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Τώρα υπάρχει εθνική στρατηγική συνεργασία αστυνομικών αρχών. Πολύ καλή ερώτηση. Ο κύριος ε, Βίτρουπ ε, βρέθηκε σε μια ευρύτερη ομάδα συνεργασίας και συντονισμού αστυνομικών δυνάμεων έγινε μία συνάντηση του IPCB σε ανώτερο επίπεδο από τον Υπουργό Ιστορικών Άτμαρ και ο Υπουργός Άτμαρ μας ε, ανέπτυξε το όραμά του ως προς τη συνεργασία με τις Αφγανικές Αστυνομικές Αρχές. Αυτή η στρατηγική δεν έχει ακόμα εγκριθεί, διότι πρέπει να περάσει από μια πολιτική διαδικασία και αναμένουμε ότι θα εγκριθεί το Μάρτιο. Μετά θα έχουμε ένα ευρύτερο, μια ευρύτερη πλαισίωση, αλλά αυτή είναι η βάση της στρατηγικής και δεν είμαστε και μόνοι μας, έχουμε πολλούς εταίρους, υπάρχει μια συνέργεια και έτσι οι δικοί μας εμπειρογνώμενες μπορούν επηρεάσουν τα πράγματα. Βεβαίως και η αμερικανική πλευρά ε, δρά πολλαπλασιαστικά στη δική μας πραγματογνωμοσύνη. Άρα και η δική του συνεισφορά είναι πολύ σημαντική. Αυτό αφορά και το ΝΑΤΟ, τη δύναμη κατάρτισης, η οποία θα κάνει αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πηγαίνει στις ε, επαρχίες για την βιωσιμότητα της αστυνομίας και για να συγκροτηθεί επιτέλους αυτή η χώρα. απαντήσω και σε ένα άλλο ερώτημα για την φιλοδοξία μας, τη συλλογική φιλοδοξία μας. Οι 400 αρκούν. Αν είχαμε περισσότερους θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά μου υπενθυμίζουν τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να είμαι ρεαλιστής. Πριν φτάσουμε τους 400, ας μην ε, τους υπερβούμε αλλά αν θέλετε μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Θα το αποδώσω στα κράτη-μέλη και θα τους πω δώστε μας ε, στέγαση και επιμελητία στις επαρχίες εκεί όπου πρέπει να επεκταθούν. Γιατί η αστυνομία δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα των κρατών μέλων πάντα. Και αυτό επιβραδύνει την όλη διαδικασία. Αν είχαμε περισσότερους θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και συνοδευτικά μέτρα. Θα ήθελα ο Κάι να μιλήσει για τις αστυνομικές δυνάμεις του Αφγανιστάν, πόσο προβάλλεται η συνεργασία, υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις. First of all, Ευχαριστώ. Βλέπετε, είδατε ήδη, καταλάβατε τι σημασία μπορεί να έχει μια σχετικά μικρή αποστολή όπως η Γιούπολ επιχείρηση. Το σημαντικότερο θα ήταν να καταλάβουμε ότι ο κυριότερος παράγοντας της επιχειρήσης του Αφγανιστάν είναι το ΝΑΤΟ και η Γιούπολ απλώς συμπληρώνει τη δράση του ΝΑΤΟ. συνδιευθύνεται από εμένα και τον Καναδό, τον Αμερικανό και έναν Ιταλό στρατηγό. Και συνεργαζόμαστε, αλληλοσυμπληρωνόμαστε και την κύρια χρηματοδότηση βέβαια την χορηγούν οι Ηνωμένε Παλιτείες. Η Ιούπολ χορηγεί την πολιτική στήριξη και είναι υπεύθυνη για την αστυνομία. Αυτό είμαι πεπισμένος ότι το θεωρούν πολύ σημαντικό και οι εταίροι, και οι μας, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ, αλλά και άλλοι. Όλοι συνεργαζόμαστε για αυτό, σε αυτό το Διεθνές Σώμα Αστυνομικού Συντονισμού και υπάρχει και μια συμβουλευτική αστυνομική ομάδα υπό έναν Καναδό όπου συνεργάζονται αστυνομικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Και αυτό είναι καλό γιατί συμμετέχουν όλοι. Το σημαντικό δεν είναι βέβαια ότι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι, αλλά ότι κινούνται όλοι προς την ίδια κατεύθυνση ο Ιταλός στο Χεράτ, ο Γερμανός στο Κανταχάρ κλπ. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε λοιπόν. Τώρα τέθηκε ένα ερώτημα για τη διαφθορά και δωροδοκία. Μήπως δεν θα έπρεπε να καταπολεμηθεί μέσω νομοθεσίας. Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Το έθεσα και εγώ στον προϊστάμενό μου στην CPCC. Δεν έχει νόημα να ζητάμε να δημιουργηθεί μια τέλεια αφγανική αστυνομία αν δεν υπάρχει το κράτος δικαίου. Υποστηρίζω λοιπόν την ιδέα για περισσότερες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς Ρωτήσατε αν βοηθούμε τους Αφγανούς. Ναι. Οτιδήποτε κάνουμε τελικά θα περάσει στους Αφγανούς. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια γερμανική, Ιρανέζικη, γαλλική αστυνομική δύναμη, αλλά αφγανική. Συγκρίσιμη όμως με τις άλλες αστυνομίες των χωρών της Κεντρικής Ασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές μας προσπάθειες έχουμε και Αφγανούς εκπαιδευτές. Χρησιμοποιούμε λοιπόν Αφγανούς και σε αυτούς θα περιέλθουν όλα αυτού τέλος. Τώρα. πώς διαχωρίζεται αυτή η εκπαίδευση μιας αστυνομίας από τις καθαρά στρατιωτικές δυνάμεις. Διαχωρίζεται, διότι εμείς θέλουμε να υπάρχει μια αστυνομία όταν θα λήξει ο πόλεμος και μετά δηλαδή. Όποτε γίνεται υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας στις εκπαιδευτικές αποστολές του ΝΑΤΟ γιατί προς το παρόν η προσπάθειά μας είναι να σταματήσουμε τον πόλεμο. Αλλά ο γενικότερος στρατηγικός μας στόχος είναι να δημιουργηθεί αυτή η μη στρατιωτική αστυνομία. Είχατε πει αν έχουμε όραμα. Ναι, έχουμε και εμείς και οι Αφγανοί έχουν να υπάρξει κάποτε ένομη τάξη και ασφάλεια στη χώρα. Κυρίως αυτό είναι το όραμα. Τώρα, αν η δική μας η Ευρωπαϊκή Αποστολή έχει αποτελέσματα σε σύγκριση με τους άλλους, μάλιστα, και οι υπόλοιποι, οι άλλοι μας σέβονται και μας υποστηρίζουν. Εξάλλου, οι συμφωνίες που υπογράφτηκαν για τις αποστολές δεν είναι μόνο μεταξύ Αμερικανών και κυβέρνηση, αλλά και Ιούπολ. Όσο για την Ευρωπαϊκή Χωροφυλακή και την συμμετοχή της στη Ιούπολ, ναι, είναι, υπάρχει και είναι πολύ σημαντική διότι αυτό που χρειάζεται είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης αφγανικής χωροφυλακής που είναι και τμήμα της στρατηγικής του Μακρίσταν. Χρειάζεται χωροφυλακή για να κρατάει τα πράγματα. Πολύ καλό πράγμα. Τώρα, αν θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και να κρατήσουμε μια αφγανική αστυνομική δύναμη, νομίζω θα μπορέσουμε γιατί ήδη αυξήσαμε τους μισθούς από 130 σε 180 δολάρια. Το μήνα, το μήνα βέβαια, 180 ταλάρια το μήνα. Και έτσι μεταξύ άλλων θα τους δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για αυτούς με τα δολάρια. Έχουν δε μπλε στολές αυτοί για να δείξουν ότι δεν είναι στρατιωτικοί, δεν έχουν χακή στολές ούτε εκείνες τις μεταμφίεσεις αλλά μπλε σκούρες μπλε για να φαίνεται ότι είναι κανονικοί αστυνομικοί χωροφύλακες και όχι στρατιωτικοί. Αλλά χρειάζεται προς στιγμή η συνεργασία με τους στρατιωτικούς. Θέλουμε όμως να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθεί μια αξιόπιστη αφγανική αστυνομική δύναμη, όχι στρατιωτική. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σοπενχάουερ. Ίσως να μην απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Μία σε μία θα ήθελα να σταθώ, γιατί είναι σημαντική. Ως προς συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, και κατά πόσο ελήψη μιας ε, συμφωνίας ασφάλειας ε, δεν υπάρχει αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο. Βεβαίως, πλήττει τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, διότι η συνεργασία in situ θα πρέπει να γίνει με βάση τη συνεργασία CPCC και των επικεφαλής αποστολής καθώς και του επικεφαλής της ε, δύναμης του ΝΑΤΟ ως προς την κατάρτιση όταν έχει δοθεί πράσινο φως. Άρα δρούμε σε μία γκρίζα ζώνη, ελπίζοντας ότι οι πολιτικές μας αρχές δεν θα δυσανασχετήσουν ως προς την έμπρακτη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, που προωθείται σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, χρειάστηκε χρόνος έως ότου η αποστολή προβάλλει ορισμένα επιτόπια μέτρα ασφαλείας. Η γραφειοκρατία έδρασε στο μεγαλείο της γιατί οι μεν δεν ήξεραν πώς να δράσουν απέναντι στους δε και δεν υπήρχε και μία πολιτική κάλυψη, δεν υπήρξε μία συμφωνία ασφαλείας και αυτό βεβαίως έχει επιπτώσει. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα ήταν καλύτερα βεβαίως να αρθεί αυτό το πολιτικό εμπόδιο. Η κυρία Άστον επεξεργαστεί και την ε, υποστηρίζω 200 τα Ως προς την ε, πρόσφατη έκθεση της Royal United Services Institute πρόκειται για ένα βρετανικό φορέα και η μελέτη διενεργήθηκε ε, με το την υπηρεσία εξωτερικής συνεργασίας στη Φιλαδέλφια. Και αυτή η μελέτη που αφορά και σχετίζεται με την συνεργασία αστυνομικών αρχών, η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε μερικές εβδομάδες πριν και αυτό που έχει σημασία είναι η μακροχρόνια μεταρρύθμιση στις αστυνομικές δυνάμεις του Αφγανιστάν. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ποιότητα, να μεταρρυθμίσουμε την αστυνομία σε μια ε, καθαρά πολιτική δύναμη, δύναμη των πολιτών, έτσι ώστε να δείτε και ποια είναι η προσθέμενη αξία της αποστολής μου. Σας ευχαριστώ και τους δύο, κύριε Κλάμπενάουερ και κύριε Βίτρουπ, για τις απαντήσεις. Ξέρω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις. Αν μπορείτε, ε, θα θέλαμε πολύ να παρευρεθείτε ε, για τη συνέχεια των εργασιών. Ο κύριος Ντέιβις, η κυρία Ντέιβις και Κάτκα θα μας μιλήσουν για την Αμερικανική στρατηγική καθώς και τις ε, δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει σε επίπεδο ασφάλειας των Αφγανικών αστυνομικών αρχών. bien. Άψογα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε. Γιατί βιαζόμαστε, βιαζόμαστε, ε? μας πιέζει ο χρόνος. Ο κύριος Ντέιβις. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να χαιρετήσω και πάλι τον κύριο Μπέρμαν και θα χαρούμε να γνωρίσουμε και άλλα μέλη της αντιπροσωπείας σας. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να χαιρετήσω και τους συναδέλφους από την ε, Ιαπωνική Αποστολή και τον Όριο Μαρουγιάμα. Τσακ, τσακ. Ε, κοιτάξτε, θα αναγκαστώ να γίνω αυστηρός άμα συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Στην ακρόαση της προηγούμενης εβδομάδας, ο γυρουσιαστής Κάρι χαρακτήρισε το Αφγανιστάν και το Πακιστάν τις πιο πολύπλοκες ε, προκλήσεις που έχουμε στην εξωτερική μας πολιτική. Και όπως ξέρετε, ο πρόεδρος Ομπάμα εξέτασε το θέμα του Αφγανιστάν και του Πακιστάν προτού ανακοινώσει την 1η Δεκεμβρίου την ε, μελλοντική πολιτική. Ήταν θετική η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και έγιναν και περαιτέρω δεσμεύσει για στρατεύματα από υπουργικό επίπεδο στο ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εταίρο κλειδί της, ε, σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν και καλωσορίζουμε την ενίσχυση των ε, σχεδίων δράση στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν και θέλουμε να ενισχυθεί η εφαρμογή και η εκτέλεση του σχεδίου αυτού. Οι διαπραγματεύσεις διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΥΠΑ συνεχίζονται και έχουν γίνει ήδη δύο προσωπικές συναντήσεις με την Βαρόνι Άστον και με τον ε, κύριο Χόλμπρουκ. Ο πρεσβευτής Άντωνι Γουέιν, συντονιστής μας ε, για θέματα οικονομικών ζητημάτων με βάση την Καμπούλ, θα καταφτάσει σήμερα στο, στις Βρυξέλλες για να διαβουλευτεί με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Κοινοβουλίου. Εν όψη του Λονδίνου ελπίζουμε ότι η Σύνοδος θα αποτύχει τέσσερα στοιχεία. Να ενισχύσει τον συντονισμό της διεθνούς αρρωγής προς το Αφγανιστάν, να ενισχύσει τις προσπάθειες του Αφγανιστάν για καλή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς τις, ε, και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, ε, πρωτοβουλίες για την επανσωμάτωση των ε, ανταρτών που επιλέγουν να ξανταχθούν στην κοινωνία και να δοθεί πλήρη αφγανική ηγεσία στο, στην αφγανική κυβέρνηση. Αυτή είναι η βασική στόχη η ενίσχυση των στρατευμάτων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ομπάμα την 1η Δεκεμβρίου έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ακριβώς τους όρους εκείνους που θα επιτρέψουν αυτή τη μετάβαση. Μετά την προηγούμενη εβδομάδα και την συνάντηση με την ύπατη εκπρόσωπο Άστον, η κυρία Κλίντον σημείωσε ότι και οι δύο πολιτικοί είναι υπέρ των στατιστικών. Η Βαρόνι Άστον είπε ότι το 50% των ε, Αφγανών είχαν υγειονομική περίθαλψη το 2002 και τώρα το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Η κυρία Κλίντο είπε ότι το 2001 ήταν ένα εκατομμύριο παιδιά παρακολουθούσαν το σχολείο. Όλα γόρια στο Αφγανιστάν. Σήμερα είναι 7 εκατομμύρια τα παιδιά αυτά, 40% των οποίων είναι κορίτσια. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα στον Αφγανιστάν. Και όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται επί τόπου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο κύριε Πρόεδρε στην Έμιλι Κάτκαρ εγώ υπηρέτησα ένα χρόνο στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ, ως ειδικό ε, επιτραμένος του πρεσβευτή. Δώσω το λόγο στην Έμιλη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Όπως είπε ο συνάδελφός μου, και εγώ πήγα επί 1,5 χρόνο στο Αφγανιστάν από τον Ιούλιο και επέτρεψα τον Ιούλιο 2009. Δεν νομίζω ότι οι τελευταίοι 6 μήνες έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Νομίζω όμως ότι μπορώ να σας πω ότι στο Αφγανιστάν, το Αφγανιστάν υπήρξε πολύ ζωτικό τμήμα τη καριέρας μου. Συνεχίζω να ασχολούμαι με τα θέματα αυτά εδώ και είναι για μένα τιμή η συνεργασία με την Ένωση που είναι σημαντικός διεθνής παράγων που συμβάλλει στις διεθνείς προσπάθειες. Πιστεύω ότι η αποστολή μας είναι αξιόπιστη. Ο πρόεδρος Ομπάμα και οι υπεύθυνοι για την εθνική ασφάλεια εκτιμούν ιδιαίτερα αυτά που κάνουμε στο Αφγανιστάν που είναι διεθνής προσπάθεια στην οποία συμμετέχει επαναλαμβάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία ξανά ευχαριστώ για τη σημαντική της συμβολή στις προσπάθειες αυτές. Διότι μόνο μέσω αυτής της διεθνούς σχέσης, εταιρικής σχέσης μπορούμε να καταλήξουμε κάποτε σε ένα ασφαλέστερο Αφγανιστάν. Όπως όλοι θα γνωρίζετε, ο πρόεδρος Ομπάμα έκανε, έβγαλε ένα σημαντικό λόγο τελευταία για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και για το Αφγανιστάν και για το Πακιστάν. Δεν ήταν κάτι το καινούργιο, αλλά βασιζόταν σε προηγούμενους λόγους και δηλώσεις και ήρθε μετά από μία μελέτη των εξελίξεων εκεί καθώς και διαβουλεύσεων με διεθνείς ε, παράγοντες και συμμάχους. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τους εξής αφέστατου στόχους στο Αφγανιστάν. Πρέπει να εκδιωχθεί από εκεί η Αλκάιντα, πρέπει οι Ταλιμπάν να μην έχουν πια τη δυνατότητα να ανατρέπουν κυβερνήσεις και ή εκλεγμένε κυβερνήσει να έχουν την εξουσία σε όλη την επικράτη. Αυτό μπορεί να γίνει με τρίτο. Πρώτο είναι η εκλελεγμένες κυβερνήσεις να έχουν την εξουσία σε όλη την επικράτεια. Αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Πρώτον, η στρατιωτική προσπάθεια που γίνεται για να αυξηθεί η δυνατότητα περισσότερη ασφάλεια του Αφγανιστάν μέσω των στρατεμάτων που έχουν ήδη αναπτυχθεί εκεί και που διασφαλίζουν την ασφάλεια ακριβώς των πολιτών. Αυτοί οι στρατιώτες θα καταλήξουν τελικά να εκπαιδεύσουν Αφγανούς αστυνομικούς και στρατιωτικούς ώστε να μπορούν από μόνοι τους να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Το δεύτερο, η συνεργασία με τους εταίρους μας στον ΟΗΕ και τον Αφγανικό λαό για να εφαρμοστεί μια πιο αποτελεσματική στρατηγική ώστε η τοπική κυβέρνηση να μπορέσει να αναλάβει από μόνη της τα καθήκοντα ασφαλείας της. Θα έχουμε πει και σήμερα ότι αυτό είναι το κλειδί, να δημιουργήσουμε μια τοπική δυνατότητα. Και τρίτον, όπως είπε η Υπουργός Κλίντον, την περασμένη εβδομάδα, η διεθνής κοινότητα έχει κάνει άλματα στις εξελίξεις για την εκπαίδευση εκεί αστυνομικών και στρατιωτών και ε, για τη δημιουργία σχολείων και χρειάζονται βέβαια ακόμη και άλλες περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως στις απομακρυσμένες υπέδρες περιοχές. Την περασμένη εβδομάδα η Υπουργό Κλίντον ε, δημοσίευσε, ανέφερε, δήλωσε μια, ένα νέο κεφάλαιο της στρατηγικής της και για όποιον ενδιαφέρεται μπορώ να σας το δώσω το έγγραφο. Πρέπει να δημιουργηθούν αφγανικοί θεσμοί για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και για να υπάρξει ένα αποτελεσματικό οικονομικό σύστημα ιδιαίτερα στη Γεωργία για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να σταματήσει η καλλιέργεια οποίου και απαρούνης και έτσι να υπάρξει μια τελείως τοπική διακυβέρνηση οι πολίτε που θα συμμετέχουν και που συμμετέχουν στα προγράμματά μα προέρχονται από όλου του τομεί. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία που έχει αυτή η πολιτική, η μη στρατιωτική πτυχή. Όχι μόνο γιατί και εγώ ήμουν μη στρατιωτικό μέλο τη αποστολής τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, αλλά και γιατί όλο και περισσότεροι συμμετέχουν Αφγανοί, όπω γεωπόνοι και άλλοι. Η Αφγανική κυβέρνηση τη χάνει επιθέσεων αυτή τη στιγμή από τους Ταλιμπάν. Σε μια μάλιστα κοινωνία που έχει καταστραφεί από έναν τριακονταετή πόλεμο. Και αυτό το λέω χωρίς να μετράμε και τα θύματα μεταξύ των αόπλων που υφίστανται επιθέσεις. Όπως αποσαφήνισε και την 1η Δεκεμβρίου ο πρόεδρος Ομπάμα, το στόχος μας είναι τι θα γίνει μετά από το πέρας της σύραξης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να υπάρξει μια σταθερή και διαρκή εταιρική σχέση με το Αφγανιστάν. Και τέλο, η τελευταία πτυχή τη στρατηγική μα είναι κάτι που δεν θα το πούμε σε λεπτομέρεια σήμερα, αλλά είναι εξίσου σημαντικό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι η επιτυχία της αποστολής μας στο Αφγανιστάν εξαρτάται ή συνδέεται και με την αποστολή μας στο Πακιστάν διότι παρά τις προσπάθειες των στρατιωτικών να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία φαίνεται ότι η Αλκάιντα έχει φωλιές στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν και από εκεί γίνονται οι επιθέσεις της κατά και των Αμερικανικών συμφερόντων. Επομένως χρειάζονται και, και πολλοί πόροι για την ενίσχυση των προσπαθειών του Πακιστάν για τον εκδημοκρατισμό του τι είναι αυτό που τα συνδέει όλα αυτά, η εταιρική σχέση, η συνεργασία της διεθνούς κοινότητας, συνδυασμένες προσπάθειες στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δυνάμεων και συνδυασμός των προσπαθειών όπως της εκπαίδευσης μιας αστυνομικής δύναμης. Ε, και φυσικά κοινό στόχο. Αν έχετε απορίες τώρα, με χαρά να σας τις λύσω. Je Ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του πρέσβη του Αφγανιστάν που θα λάβει το λόγο αργότερα. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον πρέσβη της Ιαπωνίας όπως έκανε και ο κύριος Ντέιβις και θα τον ακούσουμε διότι η συνεισφορά της Ιαπωνίας στο Αφγανιστάν είναι πολύ μεγάλη είναι ένας από τους σημαντικούς μας εταίρους η Ιαπωνία. Ο κύριος Γκάλερ ζήτησε το λόγο πρώτος. Ε, Σας ευχαριστώ. Άκουσα με ενδιαφέρον ότι ε, υπάρχουν επαφές ε, με τους Αμερικανούς και την Βαρόνια στον εδώ στις Βρυξέλλες. Να ρωτήσω και το Αφγανιστάν. Πώς θα περιγράφατε την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΙΠΑ. Πρόκειται για μια μινιμαλιστική προσέγγιση όπου απλά ενημερώνει ο καθένας τον άλλον για το τι γίνεται ή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει κάποιο, κάποιος συντονισμός, υπάρχει κάποια συμπληρωματικότητα. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα η μια αποστολή να κάνει κάτι και να το πει στην άλλη και να πει εντάξει δεν πειράζει να το κάνετε εσείς αυτό που το κάνουμε εμείς. Πώς διαμορφώνεται η συνεργασία και ταιριάζουν, συνάδουν οι δράσεις ε, και σε ό,τι αφορά τον αστυνομικό τομέα αλλά και την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους άλλους τομείς. Χαίρομαι επίσης να μιλήσω αγγλικά. για να με ακούτε και χωρίς ακουστικά. Το ερώτημα λοιπόν είναι σε ό,τι αφορά την ε, συνοπτική θεώρηση Αφγανιστάν και Πακιστάν. Άκουσα πριν από κάποιες εβδομάδες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ένα σχέδιο και για τις δύο χώρες αυτές μαζί. Δεν, ε, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Δεν μπορούμε να τις εξετάσουμε ξεχωριστά τις δύο χώρες αυτές. Ξέρουμε τι αλληλεπιδράσεις υπάρχουν μέσω των ανοιχτών συνόρων. Εσείς προβλέπετε ισχυρή συνεργασία σε τέτοια κοινή στρατηγική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ σε ό,τι αφορά την ενιαία προσέγγιση και τη των δύο χωρών. ήθελα σε αυτό το γύρο να είσαστε ιδιαίτερα συνοπτικοί στις παρεμβάσεις σας. I have a question to Emily Μία ερώτηση προς την Emily Katka. Το μόνο επιχείρημα που άκουσα τώρα ως προς τη στρατιωτική βοήθεια, την αποστολή περισσότερων στρατιωτών, είναι ότι λειτουργήσε πολύ καλά στο Ιράκ αυτό είναι συζητήσιμο, αλλά νομίζω ότι θα ήταν επικίνδυνη σύγκριση με το Ιράκ. Διότι στο Ιράκ η αντίσταση είναι κατακαιρματισμένη, δεν έχει φιλετική μορφή, βασίζεται στην πόλη, σε μια μεγάλη πόλη και σε μια επαρχία ενώ στο Αφγανιστάν υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των ε, Ταλιμπάν βασίζεται στη φιλετική, σε ένα φιλετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και έχει και, ε, έχει και τη δυνατότητα να βασιστεί στο Πακιστάν. Δεν ξέρω κατά πόσο μερικές χιλιάδες στρατιώτες μπορούν να κάνουν διαφορά. Τι διαφορά μπορούν να κάνουν σε μια χώρα που είναι 100.000 τετραγωνικό χιλιόμετρα μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Ακόμα και αν μιλάμε για μεγάλα οικονομικά κέντρα ή μεγάλες ε, πόλεις που θα πρέπει να είναι πιο ασφαλείς. Τη στιγμή που όπως, όπως έδειξαν οι επιθέσεις στην Καμπούλ την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και στην Καμπούλ δεν υπάρχει ασφάλεια. Οι επιθέσεις γίνονται έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο. Οι συμμαχικές ε, δυνάμεις μοιάζουν με δυνάμεις κατοχής. Κανείς δεν μπορεί να τις δεχτεί. Λιγότερο από όλου οι Αφγανοί. Έχουμε μεγαλύτερες ε, απώλειες σε επίπεδο αμάχων και αυτό τάσεται υπέρ των Ταλιμπάν. και οι συμμαχικές δυνάμεις ε, δεν την χάνουν υποστήριξη. Δεν βλέπω ποια λογική σας διέπει. Αυτό που βλέπω όμως είναι το άλλο τμήμα της αμερικανικής στρατηγικής, δηλαδή υποστήριξη των πολιτών. Το συζήτησα με τον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ ορισμένες εβδομάδες ε, πριν και με τον Τζον Κάρι σε ένα δείπνο Πιστεύω ότι η υποστήριξη των πολιτών θα μπορούσε να πετύχει πολύ καλύτερα χωρίς το στρατιωτικό σκέλος. Θα ήθελα την αντίδρασή σας. Ο κύριος Γκαλτιέρη. Ε, ε, ε. Ευχαριστώ. βάλω μια ερώτηση. Δεν θα ήθελα να ξαναμιλήσω για το military surge, για την ε, στρατιωτική ανάκαμψη. Μετά από τις συζητήσεις αυτής της εβδομάδας, της προηγούμενης εβδομάδας, και όπως μας υπενθύμησε ο δόκτωρ Ντέιβις, η αύξηση της στρατιωτικής δύναμης δεν είναι η μοναδική πτυχή της νέας στρατηγικής των Αμερικανών. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία από τα οποία θα ήθελα ορισμένες διασαφηνίσεις. Πώς μπορούμε να συμφιλιώσουμε τις μεν με τις δε τάσεις. Και ο Γκέιτς πρόσφατα μίλησε για την ενσωμάτωση των Ταλιμπάν αλλά υπάρχει και το δύσκολο θέμα των άλλων εθνοτικών συνιστώσεων. Διότι επλήγησαν με την πρόσφατη ετοιμιγορία του Κοινοβουλίου ως προς τον κατάλογο των Υπουργών. Και μιλάμε και για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν γενικότερα, την ε, δυναμικότητα των αστυνομικών αρχών. Δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτή την περίπτωση η ενσωμάτωση των Ταλιμπάν ή η ενσωμάτωση στοιχείων μη παστούν θα μπορούσε να βοηθήσει. Μιλάμε για μία οικοδόμηση, δημοκρατική οικοδόμηση του Αφγανιστάν. Αυτά, αυτές οι συνιστώσεις είναι συμβατές μεταξύ τους. Ο κύριος Βανμπάλ. Πρόεδρε. Πολύ ωραίος αυτός ο ήχος του κινητού. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντέιβις το εξής. Εάν θέλετε να συμμετέχουν περισσότερο οι ευρωπαϊκές χώρες στο σκέλος της ασφάλειας και στο στρατιωτικό σκέλος, Νομίζω ότι η στρατηγική των επιχειρήσεων θα πρέπει να συναποφασίζεται, όχι μόνο μερός να αποφασίζεται από τη ΣΥΠΑ. Πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία κοινή ε, συναπόφασης, δηλαδή εντός ΝΑΤΟ, με τις εμπλεκόμενες χώρες, πώς βλέπετε τη διαδικασία κοινή λήψης αποφάσεων για το μέλλον του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Ο κύριος Πετυχόφερ. Τρει ερωτήσεις έχω να κάνω. Καταρχάς, ο στρατηγός Μακρίσταλ είπε δημόσια σε αρκετές περιστάσεις ότι οι επόμενοι 12 μήνες θα καθορίσουν κατά πόσο η Δύση θα χάσει ή όχι. Τι ποσοστό αφγανικής επικράτειας δεν δέχεται επιθέσεις από τους Ταλιμπάν και ποιο θα είναι το ορόσημο τους επόμενους 12 μήνες για να πούμε ότι όχι, δεν ε, χάνουμε. Κατά δεύτερον, ποιος θα είναι ο στόχος στο μέλλον στην συνέχιση της αποστολής για την ελευθερία. Και τρίτον, πιστεύετε ότι επί του παρόντος υπάρχουν επαρκείς ικανότητες για την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους πολιτικής ασφάλειας και τι χρειαζόμαστε, θεωρείτε, για να πετύχουμε τους στόχους αυτού. Ευχαριστώ, κυρία Λούζιν. Να θέσω τις εξή ερωτήσεις. Συμφωνείτε ε, τις, με τις δηλώσεις του Ομπάμα κατά τις οποίες ε, θα υπάρχει διαρκής εμφύλιος πόλεμος στην Καμπούλ μεταξύ της Παστούν και της ε, κυβέρνησης. Αν συμφωνείτε, να πω κι εγώ αυτό που είπε ο κύριος Μπέρμαν. Η λογική συνέπεια θα ήταν η κατοχή ενός τμήματος της χώρας. Αν συνεχίσει η υποστήριξη της ε, αφγανικής κυβέρνησης όπως σήμερα. Και κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η καταπίεση του τμήματος αυτού του πληθυσμού. Μία άλλη ερώτηση που αναφέρεται και αυτή σε μελέτες των ΙΠΑ. Το 2009 σε μία μελέτη προέκυψε ότι μόνο 10% των επιθέσεων προέρχονταν από Ταλιμπάν Και σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, βασική αιτία ήταν η ανεργία, η βασική αιτία των επιθέσεων. Συμφωνείτε με την εκτίμηση αυτή. Και τελευταία ερώτηση. Ως τώρα δεν έχουμε μιλήσει ιδιαίτερα στον τύπο για θέματα λήψεων απόφασης σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν. Αλλά εσείς ποια θεωρείτε ότι θα είναι η απόφαση που θα ληφθεί. Ευχαριστώ κύριε Σκέλερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. τον κύριο Ντέιβις και την κυρία Κάτκαρ για τις παρουσιάσεις. Να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Αμερική γιατί μιλάμε για την ασφάλεια όλων μας. Και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στην, στον αγώνα αυτό. Αναφέρθηκε από τους άλλους ομιλητές ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα 5 έως 10 ετών για να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε και αναφερθήκατε και στον δεύτερο βασικό μας στόχο να ενισχύσουμε τις προσπάθειες της αφγανικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το θέμα είναι το εξής. Η εικόνα της αφγανικής κυβέρνησης και το White Rose έχουν αμαυρωθεί μετά τις τελευταίες εκλογές και αναφέρθηκαν ε, παραδείγματα αστυνομικών που κατάφεραν να αποκαλύψουν σκάνδαλα εμπορίου ναρκωτικών. Σκάνδαλα που είχαν ε, κρατηθεί κρυφά και στη συνέχεια τους κατηγόρησαν για τις αποκαλύψεις αυτές. Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι ο πρεσβευτής μπορεί να μας απαντήσει καλύτερα υπάρχει εναλλακτική στην οικονομία του οποίου και αναφερθήκατε επίσης σε διάφορα θετικά παραδείγματα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται να εξετάζουμε μεροληπτικά την κατάσταση. Είπατε ότι 85% του πληθυσμού καλύπτεται από υγειονομική περίθαλψη, ότι 7 εκατομμύρια παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία και αυτά είναι θετικά. Αλλά ο μόνος τρόπος να κερδίσουμε τον αγώνα αυτό είναι αν συμφωνήσει και ο κόσμος μαζί μας. Ευχαριστώ κυρία Κομές. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω το εξής. Αν και συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπέρμαν. Δεν συμμερίζομαι την άποψη για την νεοαπικιοκρατική στρατηγική αναφορικά με το Αφγανιστάν. Αυτό που είδα κατά την επίσκεψή μου στο Αφγανιστάν είναι αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ότι ο λαός του Αφγανιστάν ήθελε να υποστηρίξει την ε, διεθνή αυτή παρέμβαση. Γιατί έχουν δει ποια είναι τα πλέον εκτήματα, έχουν δει ποιες είναι οι βελτιώσεις, ιδιαίτερα στην, ε, σε θέματα περίταλψης και εκπαίδευσης. Αλλά ο κόσμος φοβάται, γιατί οι πιο μεγάλοι εγκληματίες πήραν θέση στην κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο, και αυτό πάει στραβά. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι συμφωνώ με τη στρατηγική που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ομπάμα και που ακολουθούν οι για την εστίαση στις πολιτικές δυνάμεις. Και ρωτώ, καταρχάς, σε ό,τι αφορά θέματα διακυβέρνησης, Ποια είναι η άποψή σας, πού θεωρείτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρόεδρο Καζά για να πετύχει αποτελέσματα και τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε α, αμέτωχοι τους εγκληματίες που παίρνουν θέσεις πολιτικές, όπως για παράδειγμα ο αδερφός του που είναι βαρόνος των ναρκωτικών. Δεν αφορά μόνο τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά και το αίσθημα της ατιμορρησίας που επικρατεί. Μετά υπάρχει και το θέμα της συμμετοχής των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Λάβαμε πολλές διαμαρτυρίες για διεθνείς και εθνικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ενώ θα έπρεπε να αποτελούν τα μέσα για να επιτευχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης, της πολιτικής ικανότητας και των κοινωνικών εξελίξεων, ουσιαστικά αγνοούνται, παραμελούνται. Πολλά χρήματα πηγαίνουν στα PRTs, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά και τα PRTs στις ε, περιοχές όπου υπάρχουν ε, και επικρατούν εξαιρετικά ανασφαλείς ε, συνθήκες, αλλά αν σε άλλους τομείς και σε άλλες περιοχές μπορούν να δράσουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις, θα πρέπει να έχουν τα μέσα για να το πράξουν. Και η λογική του ΝΑΤΟ μέχρι πριν από ένα έτος ήταν PRTs και πάλι PRTs. Λες και αυτό τώρα είναι πανάκια. Και προφανώς δεν ήταν πανάκια. Γιατί μιλάμε και για άτομα τα οποία δεν είχαν καθόλου εμπειρία επιτόπου και μιλάμε και συγκρίνουμε τα άτομα αυτά με μη κυβερνητικέ οργανώσεις με μακροχρόνια εμπειρία. Άλλη μια ερώτηση για το δικαστικό, για τη δικαστική εξουσία. Θα αποτύχουμε αν δεν επενδύσουμε και στο δικό, δικαστικό σώμα, όπως και στην αστυνομία. Μιλάμε για την οικοδόμηση ασφαλών συνθήκων και μιλάμε για έργο χρόνων για την αστυνομία αναφέρεται ότι θα χρειαστούν 10 χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα πολύ παραπάνω. Αυτό μας απασχολεί και εμάς ως Ευρωπαίους, ίσως και πιο πολύ από του τους Αμερικανούς, γιατί αφορά και την δική ασφάλεια. Και τέλος, ό,τι αφορά μια ενιαία στρατηγική για το Αφγανιστάν. Ποιο θεωρείται ότι είναι ο σύνδεσμο, ποια είναι η σχέση με την Ινδία. Δεν μπορούμε να γνωρούμε τη σχέση με το Κασμίρ. μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση του Πακιστάν. Ευχαριστούμε κύριο Ντέιβις και κυρία Κάτα στη συνέχεια. It's clear that, um... πολλά χρόνια. 5 με 10 αναφέρθηκαν ε, ως ρεαλιστικό στόχος γι' αυτό και ο Εξωτερικών τόνισε για τη συνεχή μας δράση και δέσμευση στο Αφγανιστάν μέσω διπλωματίας, μέσω οικονομικής συνδρομής και αρρωγής. Αυτό είναι ένα μακροχρόνιο σχέδιο σε σχέση με το Αφγανιστάν ως προς το θέμα της στρατιωτικής ανάκαμψης και τη σύγκριση με το Ιράκ. Νομίζω ότι έχουμε μία εκτενή προσέγγιση του, ε, ως προς το Αφγανιστάν. Αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να μπορέσουμε να κτίσουμε να οδηγήσουμε στην ανάκαμψη χρειάζονται 30.000 στρατιωτικοί επιπροσθέτως έτσι ώστε να βοηθήσουμε το πολιτικό σκέλος για την πλέον μακροχρόνια εργασία. Είναι ένα στίχημα και έχουμε αναλάβει και στο παρελθόν μαθαίνουμε από την πείρα μας αλλού και πιστεύουμε ότι σε αυτή την ε, ολιστική προσέγγιση υπάρχει προστασία του πολιτικού σκέλους, των πολιτών δηλαδή, και αυτό ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος την 1η Δεκεμβρίου σε σχέση με τις ε, συντονισμένες προσπάθειες από στρατιωτικής πλευράς. Ο συντονισμός θα γίνει στο ΝΑΤΟ μέσω ISEF και ως προς τις άλλες πτυχές συντονισμού θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Άρχισε ήδη η συνεργασία στο ε, Λονδίνο μεταξύ Άστον Κλίντον σε υψηλό επίπεδο και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα θα πρόκειται για μια προσπάθεια συντονισμού διεθνούς αρρωγής έτσι ώστε να επανενσωματωθούν και οι Ταλιμπάν, πράγμα το οποίο είναι ένα ζήτημα ουσίας, καθώς θα μας απασχολήσει και η, η πτυχή της ασφάλειας, μετάβαση του σκέλους της ασφάλειας τους ίδιους τους Αφγανούς. Τι επιθυμούν οι ίδιοι οι Αφγανοί θα δώσουμε το λόγο στον πρέσβη του Αφγανιστάν, εκείνος θα μας απαντήσει. Έγιναν ορισμένες ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει βεβαίως να δει κανείς πώς διενεργήθηκαν, πώς ερμηνεύονται, πώς τίθενται τα ερωτήματα, αλλά υπάρχουν ε, θετικά σημάδια. Οι Αφγανοί θεωρούν ότι τα πράγματα κινούνται, αρχίζουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει αρκετά και μελλοντικά. Ετέθηκε ένα ερώτημα ε, για μια εναλλακτική πορεία, διότι η ανεργία οδηγεί τους Αφγανούς στην αγκαλιά των Ταλιμπάν που μπορούν να, να τους χρηματοδοτήσουν πολύ περισσότερο σε μηνιαία βάση σε σχέση με, άλλη, με άλλη απασχόληση. Και γι' αυτό ο ειδικό απεσταλμένος, ο κύριος Χόλμπρουκ, τόνισε την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους Αφγανούς. Έτσι ώστε να μην προσχωρήσουν ούτε στους Αλιμπάν ούτε στα ναρκωτικά. Και θα σταματήσω εδώ. Ο συνάδελφος ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα, αλλά θα ήθελα να σταθώ στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ, γιατί αυτή είναι και η εργασία μου εδώ στις Βρυξέλλες. Γιατί η Ουάσιγκτον και η ΕΠΑ προσδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτή τη συνεργασία. Έχουμε υψηλούς εκπροσώπους που προσέχονται στις Βρυξέλλες για να μάθουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, διότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη ΣΥΠΑ. Ο κύριος Ντέιβις μίλησε για συντονισμό σε υψηλό επίπεδο. Επίσης ε, υπάρχει συνεργασία μεταξύ ειδικών εκπροσώπων στο Αφγανιστάν και Πακιστάν, όπως στην περίπτωση Χόλμπρουκ και ο πρέσβης, ο κύριος ε, Χολμπρουκ ήταν εδώ όταν αποτάνθηκε ο πρόεδρος Ομπάμα στο West Point στους στρατιωτικούς για την στρατηγική αυτή. Ως προς μια κοινή στρατηγική, νομίζω το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ευπρόσδεκτο από τις ΗΠΑ και μίλησα για το σχέδιο υπέρ των πολιτών η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τους ίδιους μείζονες στόχους. Μιλάμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ε, ενδυνάμωση της γεωργίας, την κατάρτιση των αστυνομικών. Έχει σημασία τι κάνουμε, πώς το προωθούμε. Όλα αυτά ορίζονται από τη βάση. Υπάρχει πολύ καλός συντονισμός και στην Καμπούλ και στο Ισλαμαμπάντ. Η διακυβέρνηση είναι ύψης τη σημασίας. Μιλήσαμε και για κατάρτιση των αστυνομικών αρχών, αλλά μιλήσαμε και για τη διακυβέρνηση την, κατά την 1η Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος Ομπάμα το τόνισε αυτό. Μίλησε για συνεργασία ε, από τη βάση προς ε, την κορυφή της πυραμίδας και οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφγανιστάν και ΕΠΑ θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους, χρειάζεται κοινή θέληση. Όσον αφορά το δικαιοδοτικό τομέα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, εντάσσονται στον ιστό υπεράσπισης των πολιτών ασχολούμαστε με θέματα ε, λεπτομέρειας σε σχέση με τη Γενική Εισαγγελία, το δικαιοδοτικό σύστημα κλπ. Πρόκειται για ένα έγγραφο 40 σελίδων. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό μας απασχολεί και η απασχόληση των πολιτών. Δεν πρόκειται μια στρατιωτική στρατηγική, αλλά για μια πολιτική στρατηγική. Ο κύριος ε, Ντέιβις μίλησε για τους στόχους ασφαλείας. Θα το αφήσω κατά μέρος, εκτός και αν ανακύψουν άλλες ερωτήσεις. Ως προς τις μη κυβερνητικέ, ε, εμείς συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους και εάν δείτε πώς οι ΙΠΑ προωθούν το όλο ζήτημα, προβάλλουμε συνεργασία με αφγανικούς φορείς για να γνωρίσουμε in situ τους ανθρώπους όχι δηλαδή ε, μόνο την κυβέρνηση αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχουμε μία ώρα με δύο παρεμβάσεις, τον πρέσβη του Αφγανιστάν καταρχήν. Θα ήθελα λοιπόν να μην ε, ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Δύο ομιλητές ζητούν το λόγο, ο κύριος Σέλερ και ο ganz θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση και να πω εξ αρχής, προκειμένου να μην ενταχθεί σε λάθος πλαίσιο, ότι οι κοινέ προσπάθειες που καταβάλλονται στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, αλλά πρακτικά από το κρατήδιό μου προέρχονται πολλοί από τους Γερμανούς αστυνομικούς που έχουν διατεθεί για την αποστολή αυτή και εγώ ήμουνα και κατά την ε, αναχώρησή τους και θα είναι και κατά την άφηξή τους. Ε, αναφέρουν ότι είναι τόσο δύσκολο για να επανδρωθεί η αστυνομία η τοπική επειδή δεν υπάρχει καμία συνεργασία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των αστυνομικών. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα των όσων ε, κάνουν οι Αμερικανοί, οι Αμερικανικές δυνάμεις και οι ιδιωτικέ δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ λίγοι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την ε, εκπαίδευση και έχουν συνήθως σχέσεις με τις τοπικές αρχές, όχι με τον κόσμο επιτόπου. Δεν ασκώ κριτικής, γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένα φιλοσοφία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Αλλά η διαφορά μεταξύ του, τι είναι ένας αστυνομικός ε, σε φιλοσοφικό επίπεδο είναι πολύ μεγάλη και σε ό,τι αφορά το έργο της αστυνομικής ε, δύναμης στο Αφγανιστάν. Μία συγκεκριμένη ερώτηση. Στην Ευρώπη υπάρχει μια αστυνομική μονάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ΗΠΑ. Υπάρχουν αυτές οι δομές. Δεν θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες δομές προκειμένου να υπάρχει πρακτικά μια στρατηγική γιατί ως προς το, προς το παρόν έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις και διάφορες φιλοσοφίες. Έχουμε και τις ε, δομές των χωρών που αποστέλνουν τις δυνάμεις και όλα αυτά συνδυάζονται δύσκολα μεταξύ τους. Ο κύριος Μπουτικόφερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζήτησα, μάλλον έθεσα τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καμία από τις ερωτήσεις μου όμως δεν απαντήθηκε. Δεν είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα κάνατε και στο Κογκρέσο. Ας υποθέσουμε ότι είσαστε στο Κογκρέσο. Απαντήστε τις ερωτήσεις μου. Πρώτη ερώτηση για το κατά πόσο έχουμε επαρκείς ικανότητες εκπαίδευσης για την αστυνομία. Δεύτερη ερώτηση για το ορόσημο, το benchmark στις επόμενους 12 μήνες για το πότε δεν θα έχουμε χάσει και για τον μελλοντικό σκοπό της αποστολής. Ευχαριστώ. εντυπωσιάστηκα από την έκκληση της Επιτροπής να υπάρξει μια ενιαία αστυνομική δύναμη στο Αφουγανιστάν. Αυτό είναι το όραμα το οποίο συμμεριζόμαστε όλοι. Να συνδυαστεί έτσι η εκπαίδευση ώστε να υπάρξει τελικά μία ενιαία αστυνομική δύναμη με την ίδια δεοντολογία, δυνατότητα και εκπαίδευση και δυνατότητες ε, κίνησης μέσα σε ολόκληρο το Αφγανιστάν. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με την αστυνομική εκπαίδευση που αναφέρατε, το σημειώνω όμως και μπορώ να σας πω ότι κάτι που μας εντυπωσίασε με τον Επίτροπο Βίντρο όταν πήγαμε για πρώτη φορά στο Αφγανιστάν το 2008 ήταν ότι είπε ότι ήθελε όσο στενότερη συνεργασία γινόταν με τους Αμερικανούς. Αυτό το θεωρήσαμε εξαιρετική πρωτοβουλία. Και είναι νομίζω ένα πρόβλημα διαφορετικών ηθών και συνηθιών εκπαίδευσης αστυνομικών, αλλά προσπαθούμε καθημερινά να τα συνδυάσουμε για να υπάρχει μια πιο συνεπής προσέγγιση, πιο συνδυασμένη. Εμείς ενθαρρύνουμε την ευπόλ στο Αφγανιστάν. Όσο για αυτά που είπατε, που ήταν όντως πολύ συγκεκριμένα, ζητώ συγγνώμη που ξέχασα να απαντήσω. Οι ερωτήσεις αυτές βέβαια θα ήταν καλύτερο να απαντηθούν από τους στρατιωτικούς συναδέλφους μας στο ΝΑΤΟ και τα είπα. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορώ να σας πω, είμαι σε θέση να σας πω τι ποσοστό υποχώρησης των Ταλιμπάν θεωρεί, θα θεωρούνταν επιτυχία. Όσο για τη συνέχιση των προσπαθειών μετά τη σύραξη, και αυτό οι στρατιωτικοί μπορούν να το απαντήσουν καλύτερα. αν έχουμε αρκετές δυνατότητες αστυνομικής εκπαίδευσης, ε, πάντα χρειάζονται περισσότερες φυσικά όσες και να έχουμε. καθώς και για τον δικαστικό τομέα χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες και προσωπικό. Είναι θέμα διαχείρισης, διαφθοράς, δωροδοκίας, όλων αυτών. Και το, το παλεύουμε, αλλά θα χρειαστούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από τους στρατιωτικούς που διαθέτουμε. Να συνδυάσω αυτά που τα λεπτά Μιλάμε για 30 πρόσθετες χιλιάδες. Ένα τμήμα τους θα είναι για την εκπαίδευση αστυνομικών. Και αυτό αναγνωρίζει το γεγονός ότι η διαχειριζόμενες και αστυνομευόμενες περιοχές είναι κάτι που πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρέσβη, σοχότατε δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Για πρώτη φορά έρχομαι εδώ στην υποεπιτροπή σας και θα ήθελα γι' αυτό να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Πρόεδρο και τους συναδέλφους που με καλέσατε να μιλήσω για την κατάσταση στο Αφιχανιστάν. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το σημαντικό ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν για τον εκδημοκρατισμό και την σταθεροποίηση της χώρας. Θα αρχίσω εκφράζοντας τις, ε, τα καλύτερες μου ευχές για το νέο έτος που ελπίζω να καταλήξει σε ευημερία και ειρήνη παγκοσμίω και διεθνώς. Το πρώτο μέρος της συζήτησης, στο πρώτο μέρος ήρθαν οι υπεύθυνοι των ε, αστυνομικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Καταρχήν, ο ρόλος της ΕΦΠΟΛ είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον η αστυνομία είναι αυτή τη στιγμή ο αδύνατος κρίκος των δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν. Χρειάζεται όντως ενδυνάμωση των δυνατοτήτων επάνδρωσης και εκπαίδευσης. 278 αστυνομικοί αξιωματικοί της αστυνομίας και εμπειρογνώμονες υπάρχουν εκεί ως εκπαιδευτές και τους ενθαρρύνουμε την Ευρώπη να αυξήσει ακόμη περισσότερο τους αριθμούς τους. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που ανέλαβε το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ φάνηκε ότι ο κόσμος έχει πιο θετική στάση ως προς την αστυνομία στο Αφγανιστάν από ό,τι προηγουμένως και αυτό οφείλεται πολύ στη διεθνή προσπάθεια. Επίσης εκτιμούμε ιδιαίτερε προσπάθειες των ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ στον τομέα της αστυνόμευσης ε, και την γερμανική συμβολή. Ο τελευταίος χρόνος ήταν ιδιαίτερα δύσκολος για το Αφγανιστάν και για τη διεθνή κοινότητα που ζει σε αυτό. Οι εκλογές ήταν δύσκολες, η ε, κατάσταση ως προς την ασφάλεια επίσης και ακούστηκαν αμφιλεγόμενα πράγματα ως προς την επιτυχία των διεθνών επιχειρήσεων που ορισμένοι είπαν ότι κατέληξαν στην αύξηση της βίας. Το 2009 ήταν το δολοφονικότερο έτος για τους αόπλους, για τους αμάχους. Αύξηση κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος των δολοφονιών. Οι Ταλεμπάν και η Αλκάιντα δολοφόνησαν δύο φορές περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οι διεθνείς δυνάμεις. 70% δολοφονήθηκαν από καμικάζι και ρασιτεχνικές βόμβες. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 45%. Αντίθετα, ένα τέταρτο των απολειών, 596 άτομα δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους λόγω των επιχειρήσεων της αφγανικής και διεθνούς δύναμης. Δυστυχώς το 2009 υπήρξε επίσης το δολοφονικότερο και για τη διεθνή δύναμη που καταπολεμεί την πληγή της τρομοκρατίας. 500, 500 περίπου θύματα της Διεθνούς Δύναμης και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα θύματα αυτά. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις θυσίες των στρατιωτών σας για την προάσπιση της υπόθεσης, της δημοκρατίας και της ειρήνευσης. Υπάρχουν τρεις λόγοι για την αύξηση της βίας σε ορισμένες περιοχές του Αφγανιστάν. Καταρχήν είναι δύσκολο να κατανικήσει κανείς την τρομοκρατία όσο υπάρχουν κέντρα του εκτός της χώρας η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο μέσα στο Αφγανιστάν. Δεν αρκεί για να εκμηδενήσει τις δυνάμεις του. Δεύτερον, το πρόβλημα της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν έχει αυξηθεί και έγινε πολυπλοκότερο παρά ποτέ. Γιατί και η σύνθεση των τρομοκρατών είναι διεθνής. Και υπάρχουν προστάτες τους εκτός της χώρας που περνούν από το Αφγανιστάν του οποίου είναι διάτρητα τα σύνορα ως γνωστόν. Και τρίτον, παρατηρήσαμε ότι οι τρομοκράτε προόδευσαν πολύ. Έχουν καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερο υλικό και καλύτερη τακτική με καλύτερο συντονισμό. Αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις διεθνείς και αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Γι' αυτό στόχος τους είναι να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό των μεγάλων πόλεων και των κομοπόλεων. Χρησιμοποιούν τις γνωστές τακτικές όπως τους καμικάζει και τις ερασιτεχνικές βόμβες, όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού και στους κυριότερους άξονες κυκλοφορίας. Είμαστε πεπισμένοι ότι το 2010 θα είναι καλύτερο από το 2009 για τρεις λόγους πάλι. Πρώτον, η διεθνής κοινότητα προσέχει ιδιαίτερα την περιφερειακή διάσταση του φαινομένου και τη ρίζα του φαινομένου, δηλαδή τις φωλιές της τρομοκρατίας, τα άσυλα. Δεύτερον, και οι αρχές του Πακιστάν δείχνουν μεγαλύτερο πνεύμα συνεργασίας με τις διεθνείς και αφγανικές δυνάμεις για την καταπολέμηση των Πακιστανών Ταλιμπάν. Είναι όμως ενισχυτικό ότι ορισμένοι κύκλοι συνεχίζουν να τους προστατεύουν, ιδιαίτερα σε βορειοδυτικές περιοχές του Πακιστάν και τις βορειοανατολικές του Αφγανιστάν. Πάντως η κυβέρνηση του Πακιστάν τον τελευταίο χρόνο έκανε πολύ περισσότερες προσπάθειες από ό,τι πριν. Ελπίζουμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές και να πολλαπλασιαστούν για να καταπολεμηθεί επιτέλους η πληγή αυτή των Ταλιμπάν στο Πακιστάν. Και τρίτον είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η διεθνής κοινότητα εκφράζει τη θέλησή της να βοηθήσει και μη στρατιωτικά για την ανάπτυξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σημαντικά τη βοήθειά τους. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι θα εφαρμόσουν μια νέα στρατηγική ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. 5 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια και άλλες χώρες φίλες επίσης ανακοίνωσαν ότι θα εφαρμόσουν νέα σχέδια. Πρέπει να δημιουργηθούν νέες σχέσεις μεταξύ ασφαλείας και ανάπτυξης, γιατί το ένα υποβοηθά το άλλο. Γι' αυτό βέβαια χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό των προσπαθειών μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ και του Αφγανιστάν. Κύριε Πρόεδρε, ορισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει στην εντύπωση ότι τα πράγματα είναι τελείως χάλια στο Αφγανιστάν. Στην Καμπούλ τελευταία έγινε μια επίθεση όπου υπήρχαν πάνω από 10 επιτιθέμενοι και υπήρξαν αρκετά θύματα και από αυτούς και από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σίγουρα έχει γεωτερέψει η κατάσταση, ιδίως προς τα σύνορα και σε ορισμένους κύριους άξονες, αλλά το περισσότερο τμήμα της χώρας είναι σχετικά ασφαλές και ήρεμο γιατί οι τρομοκράτε συγκεντρώνονται ιδιαίτερα σε ορισμένες περιφέρειες όπου είναι ιδιαίτερα μικρή η ασφάλεια. Αλλά το σύνολο της χώρας δεν υποφέρει από ανασφάλεια. Η επίθεση στην Καμπούλ μετά από μεγάλη περίοδο ηρεμίας παραμένει μεμονωμένο γεγονός και η νέα αμερικανική στρατηγική είναι ένα από τα στοιχεία που μας καθιστούν αισιόδοξου για το μέλλον. Η στρατηγική αυτή προετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις της αφγανικής κυβέρνησης και υποστηρίχθηκε από πολλούς υπουργούς εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ και από τη διεθνή κοινότητα περιλαμβάνει ουσιώδη στοιχεία για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας με κέντρο τα συμφέροντα του αφαγανικού λαού. Η νέα αυτή στρατηγική λοιπόν φροντίζει να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση για τα συμφέροντα του λαού της χώρας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μόνο με την υποστήριξη του αφγανικού λαού θα μπορέσουν οι προσπάθειες αυτές να αποδώσουν. Ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι να υπάρξει μεταφορά των ευθυνών τελικά σε Αφγανούς. Και γι' αυτό πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες, το προσωπικό των αφγανικών δυνάμεων και η νέα στρατηγική προβλέπει γι' αυτό αυξημένη προσπάθεια εκπαίδευσης και θέσεων στις δυνάμεις αυτές. Θα χρειαστεί βέβαια κάποιος χρόνος, αλλά ο τελικός στόχος είναι στόχος που τον συμμεριζόμαστε όλοι. Οι αφγανικές δυνάμεις να καταλήξουν τελικά να έχουν πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας. Μέχρι να πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός χρειάζεται να αυξηθεί η βοήθεια και η διεθνής παρουσία. Θεωρούμε λοιπόν ότι μία πρόορη απόσυρση δεν θα ήταν σωστή λύση. Κύριε Πρόεδρε, εκτός από την αύξηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και της ανασφαλείας, Άλλη αρνητική, υπάρχει και άλλο αρνητικό αποτέλεσμα που σημειώθηκε στο Αφγανιστάν όπως η αύξηση της καλλιέργειας παπαρούνης. Δυστυχώς δεν αυξήθηκε παράλληλα και ο εκδημοκρατισμός. Για τα ναρκωτικά οι αριθμοί της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών το 2009 δείχνουν ότι ο Αφγανιστάν δυστυχώς παραμένει ο κύριος παραγωγός οποίου. Ενώ έχει γίνει προσπάθεια για δεύτερο συνεχές έτος της μείωσης της καλλιέργειας. Κατά 16% περίπου μειώθηκε, ενώ οι καλλιεργούμενες επιφάνειες μειώθηκαν κατά 40%. Κατά 192.000 εκτάρια δηλαδή, έγιναν 143. Μείωση λοιπόν 35 με 40%. 37 με 40%. 20 περιφέρειες έναντι 34, σε σύνολο 34 δεν καλλιεργούν πλέον όπιον. Και η καλλιέργειά του αντιπροσωπεύει όπου υπάρχει μόνο το 2% των καλλιεργειών και μόνο σε 7 περιφέρειες νοτιοδυτικά καλλιεργείται πλέον. Σε μια ζώνη δηλαδή όπου είναι πιο δραστήριοι και οι τρομοκράτες. Το εμπόριο του οποίου αποφέρει 400 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τους Ταλεμπάν και για τους υπόλοιπους τρομοκράτες η συνεργία των Ταλιμπάν με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών αυξάνεται συνεχώς. Θα έπρεπε να τονίσουμε ότι μία από τους κύριους, ένας από τους κύριους λόγους της διαφθοράς είναι ακριβώς το χρήμα που προέρχεται από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Το 2009 ο δείκτης διαφθοράς έδειξε ότι το Αφγανιστάν είναι από τις πιο διεφθαρμένες χώρες του κόσμου μαζί με το Σουδάν. Η καταπολέμηση λοιπόν της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι ένας από τους στόχους της κυβέρνησης αλλά δυστυχώς δεν έχει ακόμη αποφέρει καρπούς. Επίσης θα έπρεπε να τονίσουμε ότι μεγάλο τμήμα των χρημάτων που δαπανά το Αφγανιστάν προέρχεται από διεθνή βοήθεια για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Στον τομέα αυτόν επίσης χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια γιατί μόνο αν βελτιωθεί η διαχείριση της χορήγησης της βοήθειας αυτής θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. Επίσης θα έπρεπε να τονίσω ότι μόνο ένα πέμπτο της διεθνούς βοηθείας περνάει από τα χέρια της αφγανικής κυβέρνησης και όλα τα υπόλοιπα από τους ίδιους τους δωρητές. Πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι το σύνολο το διαχειρίζεται η κυβέρνηση και ότι τη διαχειρίζεται επομένω τη βοήθεια άσχημα, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει και εκεί διαφθορά και δυσλειτουργία. Ορισμένοι λόγοι οφείλονται βέβαια για την κακή χρησιμοποίηση στην κυβέρνηση, άλλοι όμως όχι. Το θέμα του καλλιέργειας και λαθρεμπορίας ναρκωτικών συνδέεται με τη διαφθορά. Και ο λόγος και των δύο είναι η ανασφάλεια. Όλα αυτά ευνοούν βέβαια τις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Για να καταλήξω λοιπόν κύριε Πρόεδρε θα έλεγα ότι μπορώ να πω και κάτι αισιόδοξο παρά όλες αυτές τις προκλήσεις. Από το 2001 το Αφγανιστάν έχει κάνει προόδους σε ορισμένους τομείς όπως την υγεία, την παιδεία και την οικονομία. Χιλιάδες νοσοκομεία και σχολεία και χιλιόμετρα δρόμων έχουν οικοδομηθεί από το 2007. εκατομμύρια παιδες πηγαίνουν στο σχολείο και ένα τρίτο είναι κορίτσια, πράγμα το οποίο ήταν ε, απίστευτο με συνθήκες Ταλιμπάν. Η πρόσβαση στις βασικές υγειονομικές υπηρεσίες υπάρχει, το νόμισμα είναι σταθερό και το ΑΕΠ είναι τρεις φορές υψηλότερο από όσο επί Ταλιμπάν. Έχουμε το δημοκρατικότερο σύνταγμα της περιοχής και έχουν προβλεφθεί στόχοι που ήταν αδιανόητοι στην προηγούμενη κατάσταση. Κατά μία πρόσφατη δημοσκόπηση στο, στο BBC μεταξύ 11 και 23 Δεκεμβρίου 2009 σε ένα δείγμα 1.500 Αφγανών, το 70% των απαντήσεων δείχνει ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον. Επίσης, το 70% θεωρεί ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί το επόμενο έτος. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι τα παιδιά τους θα έχουν μια καλύτερη ζωή. Επίσης, η ανεργία καταστέλλεται. Οι Αφγανοί θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα των αστυνομικών δυνάμεων είναι καλύτερη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Μόνο το 6% τάχθηκε υπέρ μιας κυβέρνησης Ταλιμπάν. Οι περισσότεροι θεωρούν τους Ταλιμπάν ως πηγή των δεινών του Αφγανιστάν. Η μεγάλη πλειοψηφία τάσεται υπέρ της παρουσίας του ΝΑΤΟ και των ΙΠΑ στην επικράτεια. Αυτό δείχνει ότι μετά πέντε χρόνια πέντε επώδυνα χρόνια ο αφγανικός λαός στρέφεται προς, τους, προς τις χώρες φίλους όπως η ΕΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπά. Πρέπει να το τονίσουμε διότι το Αφγανιστάν θα ήθελε να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις το, κατά τα τέλη Ιανουαρίου, 28 Ιανουαρίου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις ασφαλείας και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο, στις δυνάμεις του Αφγανιστάν. Θα πρέπει να συμφιλιαθεί ο στρατός και να προωθήσουμε την καλή διακυβέρνηση και την περιφερειακή συνεργασία με βάση τις προσπάθειες και των χωρών δωρητών. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η διάσκεψη θα οδηγήσει στην ε, νέα σταθεροποίηση του Αφγανιστάν. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη για την πληρέστατη αυτή εικόνα. Θα ήθελα η Αριάν Κοντιέ να λάβει το λόγο, δημοσιογράφος σε πολλές ε, περιοχές σύραξης. Εργάστηκε στην ΑΣΕΡ, στο Αφγανιστάν και με μη θεσμικούς φορείς. Βρίσκεται πολύ κοντά στην ε, πραγματικότητα του Αφγανιστάν και δημοσίευσε και ένα βιβλίο στα γαλλικά για την κατάσταση του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η κατάσταση στο Αφγανιστάν δεν είναι καθόλου καλή και αυτό πριν από τη διάσκεψη του Λονδίνου. Οι εκλογές δεν είναι συνταγματικές, δεν είναι νόμιμες, δεν έχουμε Κυβέρνηση ουσίας, οι βουλευτικές εκλογές διενεργήθηκαν, η κατάσταση δεν είναι καλή. Όπως διαπιστώσατε, τα Ηνωμένα Έθνη το τόνισαν αυτό. Υπήρξα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ο Ρίτσαρτ Χόλμπροκ είχε μια μεγάλη διαφορά τον κύριο Καζάη, με τον πρόεδρο Καζάη και ο γερουσιαστής Κέρι επέλυσε τη διαφορά. Άρα και από πλευράς ασφάλειας δεν βαίνουν καλά τα πράγματα. Το 2007 η επανάσταση πρώτων θυρών της Καμπούλ σήμερα βρίσκεται εντός της Καμπούλ μεγάλη ε, αμφισβήτηση και πιστεύω ότι και ο αφγανικός ε, στρατός δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Αυτό το βλέπουμε πέρα από τις δημόσιες δηλώσεις ελπίδας ως προς την αστυνομία. Πολλά πρέπει να γίνουν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αστυνομία που υπηρετεί τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Η διάσκεψη του Λονδίνου θα ασχοληθεί με θέματα ασφάλειας. Η καλή διακυβέρνηση είναι ένα αναγκαίο στοιχείο. Και μην ξεχνάμε ότι οι βασικές δυνάμεις είναι αμερικανικές και ας έχει ανακοινώσει η Ευρώπη μια παρουσία 5.000 στρατιωτών. Το Λονδίνο είναι η διάσκεψη της τελευταίας ευκαιρίας για να αποσαφινιστεί η κατάσταση και ίσως και να βελτιωθεί. Και ο ρόλος της αστυνομίας θα αναφερθεί εδώ και δύο χρόνια. Η Integrity Watch Afghanistan η οργάνωση αυτή διενέργησε μια έρευνα η οποία κατέδειξε ότι η αστυνομία δεν είχε καθόλου καλή εικόνα. Ήταν πιο διεφθαρμένη, ο πιο διεφθαρμένος θεσμός μετά από τα δικαστήρια και την δικαιοσύνη. Άρα η αστυνομία είναι ο φτωχός συγγενής της ανοικοδόμησης και η UPOL μας είπε ότι δεν ήταν προτερότητα, το είναι αδιαμφισβήτητο και σήμερα έχουμε μεγάλη πορεία να διανύσουμε ακριβώς επειδή δεν έγινε μεταρρύθμιση σε επίπεδο αστυνομίας ή έγινε μία ανεπαρκής μεταρρύθμιση. Όταν διαβάσουμε τις συμφωνίες της Βόνης γίνεται έμεσα μνήμα μια μεταρρύθμιση του στρατού για να δημιουργήσουμε έναν εθνικό στρατό. Τότε τι συνέβη. Πολλοί καταπολέμησαν τους Ταλιμπάν ή της αντισοβιετικής ε, τζιχάντ και οι οποίοι κατέφυγαν στην αστυνομία ή στο Υπουργείο ε, Εσωτερικών έτσι ώστε να λειτουργήσουν με αυτά τα βακούφια και τους φύλαρχους. Έτσι ώστε να καρποθούν την κατάσταση. Ο Αχμέτ που ήταν υπουργό Εσωτερικών το 2003 που προσπάθησε να προβεί σε μεταρρύθμιση, δεν τα κατάφερε και αναρωτιόμαστε κατά πόσο και ο πρόεδρος ε, Καρζάη το επιθυμούσε αυτό ο Μαχμέτ το 2004 ζήτησε τη μεταρρύθμιση και της αστυνομίας. Αλλά δεν τα κατάφερε. Το 2006 είχαμε την επάνωδο των ε, Ταλιμπάν στο Κανταχάρ, Έλμαν. Άρα είχαμε μία αναζωπήρωση των επαναστατικών δυνάμεων και οι Αμερικανοί τι είπαν «Α, κάτι πρέπει να κάνουμε». Λέω οι Αμερικανοί γιατί αυτοί είναι οι κύριοι του παιχνιδιού, δεν είναι οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί λοιπόν, η διεθνής κοινότητα, δηλαδή οι Αμερικανοί, τι είπαν «Α, θα συνεργαστούμε με αυτό τον αδύναμο κρίκο, την ε, αστυνομία στον Νότο θα τη μεταρρυθμίσουμε. Το 2002 24 εκατομμύρια δολάρια ε, δίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το πακέτο. Και όπως γνωρίζουμε οι Αμερικανοί έχουν μία ε, στρατηγική καθαρά ε, στρατιωτικής υφής και μέσω ενός οργανισμού προσπάθησαν να μεταρρυθμίσουν την αστυνομία η οποία ε, είναι μια αστυνομία καταστολής των επαναστατικών δυνάμεων. Σήμερα λοιπόν στο Αφγανιστάν όποιες και να είναι οι προσπάθειες της EUPOL που λειτουργεί ως ε, αστυνομική δύναμη υπέρ των πολιτών, τι κάνει οποία υποστηρίζει την ISAF, ε, διότι μιλάμε για 400.000 στρατιωτικούς που χρειάζονται να λάβουν υπόψη την ε, τοπογραφία του Αφγανιστάν. Τώρα θα έχουμε περίπου 140.000 διεθνή δύναμη συν το MDS που είναι οι μυστικές υπηρεσίες του Αφγανιστάν. Άρα φτάνουμε στις 400.000 αλλά κατά των πολιτών με μια αστυνομία η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αντεπανάσταση γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε κάθε επαρχία, σε κάθε γειτονιά υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Άρα υπάρχει η ευρωπαϊκή τάση της ε, αστυνομίας υπέρ των πολιτών και απ' την άλλη υπάρχει η τάση της αστυνομίας καταστολής των ε, αντεπαναστατικών δυνάμεων. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Σήμερα λοιπόν έχουμε ποσότητα, ίσως ναι, ίσως όχι ποιότητα. Έγινε λόγος για διαφθορά και στην αστυνομία. Η αστυνομία δεν ασχολήθηκε με την ε, διαφθορά επί Ο πρόεδρος Καρζάη έπρεπε να απομακρύνει τον αδελφό του. Έπρεπε να απομακρύνει και άλλους ηθήνοντες επικεφαλής της ε, περιφέρειας του Κανταχάρ, δεν το έκανε ξεχνάμε και τη συμμετοχή των, ε, του αδελφού του Προέδρου Καρζάη στο εμπόριο ναρκωτικών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον ρόλο του, του Δημάρχου της Κανταχάρ. Και στη συνέχεια υποτίθεται ότι ο πρόεδρος Καρζάη θα καταπολεμούσε τη διαφθορά. Ο δήμαρχος όμως ε, καταδικάστηκε σε κάθυρξη τεσσάρων ετών. Ο πρόεδρος Καρζάη όμως εκφράζει την εμπιστοσύνη του προς το δήμαρχο, ο οποίος έχει εφεσιβάλει. Άρα δεν έχουμε αστυνομία υπέρ των πολιτών. Ούτε πολέμηση της διαφθοράς. Euh, Το 2007 πληρωνόταν 160 δολάρια ένας ε, ε, αστυνομικός. Συμμετείχε και στο σχήμα Dime Corps. Είναι μεγάλη νοσταλγή του πολέμου πολλές φορές, όπως είδαμε και από τη ε, δράση του στα Βαλκάνια. ιστορία της Time ε, Corps ήταν η ψηλότερη, η αμοιβή αυτού του φορέ ήταν η ψηλότερη από όλων των αστυνομικών μέσα σε ένα χρόνο. Υπάρχουν βεβαίως νησίδες ελπίδας, όπως είπε και ο πρέσβης. Οι Αφγανοί δεν αγαπούν τους Ταλιμπάν, αυτό είναι σίγουρο και είναι πολύ σημαντικό. Τους έζησαν, τους βίωσαν και τους λείπει η δικαιοσύνη πολλές φορές και η ασφάλεια που τους εξασφάλισαν οι Ταλιμπάν, αλλά δεν τους αγαπούν. Υπάρχει μία αυστηρότητα περίεργη και στρεβλωμένη αυστηρότητα που προβάλλουν οι Ταλιμπάν, δεν μπορούν ε, τα παιδιά να παίξουν με αϊτούς σε πάση περιπτώσει έχουν μια διαστραμμένη λογική. Δεν ξέρουμε βεβαίως, ε, δεν ξέρουμε ποιο σημείο ελέγχει την κατάσταση η δύναμη των Ταλιμπάν, αλλά οι Ταλιμπάν δεν κατέχουν μεγάλες πόλεις, ούτε το Κανταχάρ, ούτε τη Τζαλαλαμπάντ. Έχουν ε, υψηλή παρουσία στον ιστορικό νότο, αλλά δεν κρατούν καμία πόλη, ούτε καν τους ε, μεγάλους οδικούς άξονες. Μεταξύ Καμπούλ και Κανταχάρ είναι δύσκολη η διέλευση, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει διεθνής, υπάρχουν διεθνείς δυνάμεις και ο ανεφοδιασμός ε, δεν είναι πάντα εύκολος. Στη διάσκεψη του Λονδίνου, οι Αφγανοί και οι διεθνείς δυνάμεις θα εξεύρουν μία νέα μορφή εταιρικότητας. Θα ήταν ε, τερατώδες λάθος να πούμε ότι γυρίζουμε σελίδα για την περιοχή αλλά ίσως βρισκόμαστε στην, ε, τέλος πάντων σε μια κατάσταση όπου η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ήσασταν ένα χήμαρος, μία πλημμυρίδα και δεν μπορούσαν εύκολα να σας, να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή της ΑΦΕΤ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομα αλλά και δύσκολα ερωτήματα προς τους Αμερικανούς ε, ομολόγους μας, που είναι διπλωμάτες καριέρας. Δεν περιμένω λοιπόν πλήρης απαντήσεις, γιατί είναι πολιτικό το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Και είναι πολύ πολιτικές οι ερωτήσεις, αλλά και δύσκολες. Η πρώτη λοιπόν, για τα ναρκωτικά στο Αφγανιστάν απαντήσατε στους συναδέλφους ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε πλήρως γιατί είναι θέμα για τους ειδικού. Και το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δυστυχώς η πιο πολλή ηρωίνη που έρχεται στην Ευρώπη προέρχεται από το Αφγανιστάν, άνω του 92%. Και στη Ρωσία υπάρχει αφγανική ηρωίνη που σε 10 χρόνια κατάφερε να διεισδύσει σε δύο μεγάλες περιοχές του κόσμου. Έχει σημασία λοιπόν. Ίσως και αυτό να αποτελεί το μοναδικό λόγο για τον οποίο θα πρέπει η Ευρώπη να βρίσκεται σήμερα στον Αφγανιστάν. Όταν οι Αμερικανοί μπήκαν στην Καμπούλ, δεν υπήρχε παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν. Τότε, εκείνη τη χρονιά, οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν την ε, καλλιέργεια υπό την πίεση των Αμερικανών και κατέδειξαν ότι ήταν δυνατόν με πολιτικά μέσα, μάλλον καταδείχθηκε ότι με πολιτικά μέσα ήταν δυνατόν να απαλληφθεί η καλλιέργεια οποίου εννέα χρόνια αργότερα η καλλιέργεια του οποίου ανθεί. Ακόμα και αν υπήρξε μια μικρή πτώση τα τελευταία χρόνια. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Τι συνέβη. Τι ναι. συνέβη. Ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας γνώμη για να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορείτε να απαντήσετε. Δεύτερη ερώτηση. Σήμερα το πρωί είμαι σίγουρη ότι το διαβάσατε ε, τις δηλώσεις ε, και την συνέντευξη του στρατηγού Μακρίσταλ στους Financial Times. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιατί αν θέλει κανείς να μάθει κάτι για το Αφγανιστάν και τη σχετική πολιτική, θα πρέπει να ακούει τι λένε οι στρατηγοί και όχι τι λένε οι πολιτικοί. Γιατί είναι ξεκάθαρες οι θέσεις του και οι τοποθετήσεις του για το τι θα πρέπει να γίνει στο Αφγανιστάν. Και αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με αυτά που κηρύττουν οι, Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και ο κύριος Όλμπρουκ είπε ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε να μείνουμε στο Αφγανιστάν πιο πολύ από ότι στο Βιετνάμ. Αλλά ο στρατηγός Μακρίσταλ έχει σαφείς ιδέες και είπε δύο στοιχεία, πολύ βασικά. Καταρχάς ότι αρκετή, αρκετός αγώνας έχει δοθεί από στρατιωτικής πλευράς. Δηλαδή, και αυτό είναι σημαντικό για στρατιωτικό, ότι από στρατιωτικής πλευράς δεν θεωρεί ότι υπάρχει πολύ περιθώριο. Κατά δεύτερον, ότι λογική συνέπεια θα ήταν να περάσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ισχυρή στρατιωτική α, θέση γίνεται. Και αυτό είναι λογικό. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό όμως για μας να ξέρουμε τι περιμένετε από την διάσκεψη του Λονδίνου για τα δύο θέματα αυτά. Τι θα γίνει για την παραγωγή των ναρκωτικών επειδή σε νέα χρόνια καμία από τις δυνάμεις κατοχής δεν πέρασε στρατηγική για την καταπολέμηση και την κατάργηση της ε, παραγωγής οποίου υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο λοιπόν. Και δεύτερον, ποια η θέση σας για την συνέντευξη του στρατηγού Μακρίσταλ. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρεσβευτά, είπατε στην ε, παρουσίασή σας ότι η Αφγανική κυβέρνηση του 2009 έκανε πολλά για να πετύχει τη μείωση της υποστήριξης του κοινού προς τους Ταλιμπάν. Θα ήθελα να μας πείτε συγκεκριμένα ποια ήταν τα πιο, συγκεκριμένα, τα πιο σημαντικά μέτρα που ελήφθησαν για να μειωθεί η υποστήριξη προς τους Ταλιμπάν. Κυρίως ε, στο νότο αλλά και στον, στο βορρά αλλά και στο νότο. Σε συνεργασία με τις διεθνείς δυνάμεις και κατά δεύτερον γίνονται τέτοιες ε, σκέψεις και από την αφγανική κυβέρνηση για τις συζητήσεις με τους πιο μετριοπαθείς εισαγωγικά Ταλιμπάν και μία πιο γενική ερώτηση. Τι σημαίνει αυτός ο όρος μετριοπαθής Ταλιμπάν και να ενημερώσω την ε, Επιτροπή μας για τη χτεσινή επίθεση στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ όπου τέσσερις ε, βούλγαροι στρατιώτες ε, τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και Ρουμάνοι στρατιώτες και πολλοί συναδελφοί εδώ στο Κοινοβούλιο μάλλον κάποιοι συναδέλφοι του Κοινοβουλίου ήταν παρόντες, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Αλλά από ό,τι φαίνεται στο Αφγανιστάν πουθενά κανείς δεν είναι απόλυτα ασφαλής ακόμη. Ευχαριστώ κυρία Κόμες. Κοιτάξτε, εξετίμησα ιδιαιτέρως τις απόψεις της Δεσποινίδος Καντιέ. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η προσέγγιση κάποιου που γνωρίζει καλά τα πράγματα επιτόπου αλλά δεν εκπροσωπεί καμία από τις ε, δυνάμεις που επίσημες δυνάμεις που λειτουργούν εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι προς τον κύριο Πρέσβη και τους εκπροσώπους των ΗΠΑ της αποστολής των ΙΠΑ. Αφού μιλήσαμε για διαχείριση και διακυβέρνηση και τη στρατηγική καταπολέμηση διαφθοράς γορδοκές και ναρκωτικών, θα να πω ότι δύο προβλήματα που είδαμε πέρυσι, όποτε μας μίλησαν αντιπροσωπείες στο Αφγανιστάν εδώ, αφορούσαν τον νόμο για, τα, για την ελευθεροτυπία που δεν ήταν καθόλου δημοκρατικός και τον οικογενειακό νόμο που ακολουθούσε τους δρόμους των Ταλιμπάν χοντρικά. Υπάρχει κανένα μια πρόθεση να αλλάξουν αυτά. Ναι, κύριε Βαν Πρόεδρε. Πράγματι ο πρέσβης του Αφγανιστάν από τότε που ήμουν βουλευτής στην Ολλανδία. Ξέρω ότι πάντοτε ήταν ανοιχτό σε διάλογο και τώρα που είμαι ευρωβουλευτής ερωτώ το εξή. Οι βουλευτικές εκλογές είναι πάντα σημαντικές σε οποιαδήποτε χώρα. Αποφασίσατε να αναβληθούν. Τι λέει η κοινή γνώμη αλλά και μεταξύ πολιτικών, τι λέγεται για αυτή την αναβολή. Γιατί θα μπορούσε να θεωρηθεί ως χειραγώγηση. Μπορείτε να μου το σχολιάσετε παρακαλώ. Ο κύριος Μπούτικ Χόφερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία ερώτηση να απευθύνω προς τον κύριο Πρεσβευτή και μία ερώτηση προς την κυρία Καντιέ. Κύριε Πρεσβευτά, ο κύριος Ντέιβις προηγουμένως μίλησε και ανέφερε ότι ένας από τους στόχους της ε, διάσκεψης του Λονδίνου είναι κάποιες ε, δυνάμεις ε, επαναστατικές να ενσωματωθούν εκ νέου στην κοινωνία. Θα ήθελα να ακούσω την απόψη της δικής σας κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Είναι μερικαντελιστική αυτή η ενσωμάτωση. Να τους δώσουμε χρήματα για να σταματήσουν να μας πυροβολούν είναι πολιτική αυτή η ενσωμάτωση. Και αν είναι πολιτική, ποιους ε, καλύπτει. Αυτό που μου είπε ο στρατηγός Μακρίσταλ που αναφέρθηκε μόλις, δεν ε, χρησιμοποιεί τον όρο μετριοπαθής Ταλιμπάν και νομίζω ότι ο στρατηγός είναι αρκετά ρεαλιστικός αναφέροντας ότι θα πρέπει να μιλήσουμε, να συνομιλήσει κανείς με τον εχθρό για να πετύχει αποτελέσματα. Εσάς ποια είναι η θέση σας. Ο πρόεδρος Καρζάη έχει δώσει μεγάλη πολιτικό βάρος σε αυτή την έννοια της επανενσωμάτωσης. Αν θα μπορούσατε να διευκρινίσετε τι εννοείτε. Και μία ερώτηση λοιπόν τώρα προς την κυρία Καντιέ είπατε ότι η διάσκεψη του Λονδίνου ενδεχομένως να αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία για τη μεταστροφή στο Αφγανιστάν. Ο πρεσβευτής έδωσε σε διάφορες ε, περιπτώσεις την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο σημαντική η διάσκεψη του Λονδίνου και το σημαντική ήταν η δήλωση του Πρόεδρου Ομπάμα τον Δεκέμβριο ποιες ε, θεωρείτε, ποια θεωρείτε ότι είναι τα τρία πιο σημαντικά αποτελέσματα που θα πρέπει να πετύχει η Σύνοδος του Λονδίνου για να στεφθεί με επιτυχία. Η κυρία Λόιζανγκ, λέει ο πρόεδρος. Ε. Μιλήσαμε πολύ για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Δεν είμαι εδώ ως διπλωμάτης. Γι' αυτό και θα κάνω πιο συγκεκριμένη την ερώτησή μου. Κύριε Πριζευτά, αναφέρατε ως αιτία της ε, καλλιέργειας ναρκωτικών το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών. Ασφαλώς και χωρίς το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών δεν θα υπήρχε και το πρόβλημα αυτό και υπάρχουν διάφορα θέματα που τίθενται και από το δικό μας κόμμα σχετικά με την νομιμοποίηση ενδεχομένω των ναρκωτικών. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχουν να κάνουν με το εμπόριο, αλλά σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΟΗΕ, 75% των εσόδων από τα ναρκωτικά καταλήγουν στις τσέπες της κυβέρνησης. είναι παράλογο. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία άλλη κατεύθυνση. Κατά δεύτερον, είπατε πρεσβευτή ότι η αιτία των συγκρούσεων είναι η τρομακρατία και ότι η τρομοκρατία βρίσκεται εκτός των συνόρων της χώρας. Και συνέχεια αναφέρονται οι Ταλιμπάν. Και είπατε κι εσείς ξεκάθαρα ότι η εξουσία των Ταλιμπάν μπορεί να είναι πιο περιορισμένη. Η αιτία των συγκρούσεων δεν είναι πιο πολύ η φτώχεια στη χώρα σας και η επανάσταση αυτή που διαρκώς αναφέρατε. Είπατε ότι μεγάλο έργο της νομικής δύναμης είναι η καταπολέμηση και η κατάπνιξη των ε, εξεγέρσεων. Ποιοι είναι όμως αυτοί που εξεγείρονται, από πού προέρχονται, όλοι απ' έξω από το Αφγανιστάν έρχονται. Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Και αυτή η εξέγερση δεν προέρχεται από τους παστούν που έχουν χάσει τα δικαιώματά τους ανατολικά της χώρας και θα ήθελα κάποια αριθμητικά στοιχεία. Οι συγκρούσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και εξηγερθέντων το 2009 έφτασαν σε ένα ιστορικό ρεκόρ 16.000. Δεν ε, ήταν όλοι αυτοί τρομοκράτες που είχαν μπει στη χώρα παράνομα. Αυτό είναι παράλογο. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονα τον είπα το 2005 ε, υπήρχαν εξεγέρσεις σε 11 από τις 34 περιφέρειες, ενώ κάποια χρόνια μετά σε 33 από τις 34 περιφέρειες. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι όλα αυτά είναι από το εξωτερικό της χώρας. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι έχει βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση της ασφαλείας το 2009-2010 και κλείνοντας να πω ότι οι θετικές εξελίξεις που παρουσιάστηκαν για την αφγανική κοινωνία είναι πολύ σχετικά τα στοιχεία αυτά γιατί το 61% των Αφγανών εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αναρωτιέμαι από πού προέρχονται τα αριθμητικά στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Merci, Monsieur le Président. υποστήριξη προς τους Ταλιμπάν. Ποτέ δεν ήταν ε, δημοφιλής οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Ήρθαν με τη δύναμη των όπλων. Πολύ συχνά λέγαμε ότι το Αφγανιστάν ήταν όμοιρος ορισμένων χιλιάδων ε, ένοπλων. Η Ταλιμπάν ήταν μία από αυτές τις ομάδες που ε, έπιασε το Αφγανιστάν σε ομοιρία και το Αφγανιστάν απέρριψε την κυβέρνηση Ταλιμπάν. Είχε μια υποστήριξη της τάξης του 5-6%. Ως προς τους μετριοπαθείς ε, Ταλιμπάν. Σας είπα ότι το κατακεφαλή εισόδημα τριπλασιάστηκε μετά το 2001. Γιατί ήταν 180 δολάρια το 2001. Σήμερα είναι 450 δολάρια το κατακεφαλή εισόδημα. Άρα η χώρα είναι πολύ φτωχή. Και πολύ ε, βρίσκονται στο πλευρό των Ταλιμπάν εξαιτία της φτώχειας. Διότι οι Ταλιμπάν είναι πολύ πιο πλούσιοι από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν πληρώνουν τρεις-τέσσερις φορές πιο πάνω από την κυβέρνηση Αφγανιστάν. Η φτώχεια λοιπόν υποχρεώνει μερικούς να ε, συμμετέχουν, να υποστηρίζουν τους Ταλιμπάν. Εδώ μιλώ για τις στρατιωτικές δυνάμεις. Γι' αυτό ζητάμε και αναπτυξιακά προγράμματα για να υπάρχει ασφάλεια και στο Νότο και προς Ανατολάς, έτσι ώστε να δώσουμε εργασία σε αυτούς τους φτωχούς, έτσι ώστε να μην εργάζονται για τους Ταλιμπάν, οι οποίοι ε, σφαγιάζουν αθώους. Διακυβέρνηση. Συμφωνώ ότι η διακυβέρνηση είναι καθόλου καλή αλλά αν δούμε το Αφγανιστάν σήμερα και δούμε την κατάσταση από πλευράς Αμερικής ή Ευρώπης, η κατάσταση είναι δραματική. Αν δούμε την ιστορία του Αφγανιστάν, το 2001 δεν υπήρχε κυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Το 2001 δεν υπήρχε νομοθετική εξουσία δικαιοδοτική, δεν υπήρχε εθνικό στρατός, δεν υπήρχε εθνική αστυνομία. Έκτοτε προόδευσε το Αφγανιστάν, ακόμα και στην τομέα της διακυβέρνησης. Σήμερα έχουμε τις τρεις εξουσίες που προαναφέραμε. Και θα πρέπει αξιολογήσουμε και το γεγονός ότι η εκτελεστική εξουσία απέρριψε το ίμιση των Υπουργικών Χαρτοφυλακίων. Μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε τον δεσποτισμό που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Τώρα το Αφγανιστάν έχει μια κυβέρνηση. 14 υπουργοί εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο. Έχουμε τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υφίσταται κυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Εγώ ως Αφγανός εκτίμησα το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συζητά ορισμένα ζήτηματα με την κυβέρνηση και απορρίπτει και μερικούς υπουργούς ως προς τον νόμο της οικογένειας. Μιλάτε για τον Σιητικό νόμο. Ο Σιητικός νόμος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και μετά κοινοποιήθηκε και από την, τον Πρόεδρο. Αλλά ο Πρόεδρος ζήτησε την αναθεώρηση του νόμου και αναθεωρήθηκε ο νόμος. Και οι περισσότερες ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις, ακόμα και η ανθρωπιστική οργάνωση του Αφγανιστάν που είναι τόσο επικριτική, είπε ότι τώρα ο νόμος καλώς έχει. Το Αφγανιστάν απαρτίζεται κατά 20% από ΣΥΙΤΕΣ. Αυτό το μέρος του πληθυσμού επισκιάζεται από τους Σουνίτες και για πρώτη φορά στην ιστορία του Αφγανιστάν δίδονται ορισμένα δικαιώματα και, για τους, ε, και στους ΣΥΙΤΕΣ, ιδιαίτερα στον τομέα της οικογένειας. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδος. Με βάση το νέο σύνταγμα. Δηλαδή οι ΣΥΙΤΕΣ έχουν δικαιώματα στον ε, τομέα της, ε, του οικογενειακού δικαίου. Τώρα ο νόμος έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί. Η κοινωνία του Αφγανιστάν είναι πολύ παραδοσιακή. Ζήσαμε τη δημοκρατία τρεις φορές. Το 19 μετά την ανεξαρτησία του Αφγανιστάν, τότε ο βασιλιάς προέβη στη σύσταση ενός κοινοβουλίου, αλλά προχώρησε πολύ γρήγορα. Μετά η παραδοσιακοί εναντιώθηκαν και ο βασιλέας εγκατέλειψε τη χώρα. Το 1963 ήταν η δεύτερη μας εμπειρία. Ίσως είχαμε την καλύτερη, το καλύτερο σύνταγμα της Ασίας εκείνη την εποχή. Δηλαδή είχαμε μια πραγματική δημοκρατία η οποία μεσουράνησε στο Αφγανιστάν. Υπήρχε ελευθερία του εκφράζεστε. Και όλα έληξαν με εξωτερική παρέμβαση. Έκτοτε, το 78, μετά το 78, το Αφγανιστάν βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση μέχρι το 2001. τους βρισκόταν υπό έλεγχο στρατιωτικών δυνάμεων. Το 2001 για πρώτη φορά είδαμε ότι ο πληθυσμός έζησε μία μεγάλη περίοδο ελπίδας. Οι προσδοκίες βεβαίως του λαού ήταν πολύ υψηλότερες από αυτό που πραγματώθηκε. Και γι' αυτό πολλοί απογοητεύτηκαν. Και για τέσσερα χρόνια Όλες οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο πληθυσμός δεν υποστήριζε αυτή τη διαδικασία. Φέτος ε, για πρώτη φορά βλέπουμε μία αλλαγή. Δηλαδή ο αφγανικός λαός γίνεται πιο αισιόδοξο για το μέλλον της χώρας και δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την συνέχεια αυτής της διαδικασίας, εκδημοκρατισμός, ανοικοδόμηση και ούτω καθεξής. Έχετε όμως δίκιο, το πρωταρχικό πρόβλημα του Αφγανιστάν είναι το θέμα της φτώχειας. Εάν οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν τη φτώχεια, τη χρησιμοποιούν και οι άλλοι, διότι η φτώχεια είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη μάστιγα στο Αφγανιστάν. για τις βουλευτικές τώρα εκλογές. Εάν το Αφγανιστάν διοργανώσει βουλευτικές εκλογές στις ε, προθεσμίες που προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή το Μάιο, όλοι το επικρίνουν. Πώς ε, σε μια χώρα που δεν υπάρχει ασφάλεια θα διενεργηθούν εκλογές. Διότι από το Σύνταγμα προβλέπεται η ημερομηνία ε, διενέργειας εκλογών. Αλλά αν δεν υπάρχει ασφάλεια, αν δεν μπορεί ο πληθυσμός να ψηφίσει σωστά, δεν θα είναι καθόλου εύκολο, όπως ίσχυσε και με τις προεδρικές εκλογές. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει καθολικότητα, γι' αυτό έγινε αναβολή για τέσσερις μήνες. Τέσσερις μήνες δεν είναι και πολύ. Έτσι ώστε οι εκλογές να διενεργηθούν ε, υπό το κατάλληλο κλίμα. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη, η Αριάν, για το ερώτημα που σας... Ναι, πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Τρία έπρεπε να προκύψουν, έπρεπε να προκύψουν από τη διάσκεψη του Λονδίνου. Δηλαδή, ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, δεν πρέπει να κρυβόμαστε και στρατιωτικά και πολιτικά και αναπτυξιακά. Και η κατάσταση αυτή κρατάει 8 χρόνια και συνεχώς χειροτερεύει. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια φάση όπου αν δεν κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε μια σοβαρή εταιρική σχέση στην πράξη με τη διεθνή κοινότητα και με τους στρατιωτικούς διότι οι στρατιωτικοί δεν πρόκειται να καταλήξουν σε καμία νίκη παρά μόνο αν συνοδευτεί η δράση τους με την καλή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη. Επομένως, καταλήγω ότι αυτό φάνηκε τα τελευταία 8 χρόνια και ως προς την σύραξη νομίζω ότι ναι μεν οφείλεται και στη φτώχεια αλλά όχι μόνο. Θυμηθείτε τις αγροτικές επαναστάσεις στο Μεσαίωνα, όπου έβγαιναν οι αγρότες με τις τσουγκράνες και ήθελαν να ρίξουν την κυβέρνηση. Ναι, εντάξει, υπάρχει η παρέμβαση του Πακιστάν, υπάρχουν οι φανατικοί της Αλκάιντα, αλλά πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και λόγια λόγους δικαιοσύνης και όχι μόνο φτώχειας. Ο κύριος Ντέιβις. Θα αφήσω τη συνάδελφο. Να απαντήσω για τα ανακαλυτικά. Επειδή ήμουν στο Αφγανιστάν το 2008 και 2009 και μπορεί να μην μπορώ να απαντήσω το, στο γιατί αυξήθηκε η καλλιέργεια της παπαρούνας, αλλά να πω ότι όταν ξεκίνησε την θητεία του πρόεδρος ο Ομπάμα και ο πρεσβευτής Χολμπρουκ είπε ότι προφανώς η στρατηγική για τα ναρκωτικά στο Αφγανιστάν δεν λειτουργούσε. Και κάποια από τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται τώρα και τα οποία οι ΙΠΑ εξετάζουν περιλαμβάνουν και την εξέταση των αιτιών. Όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές ροές προσθέτοντας ε, επιπλέον προσωπικό στην εξέταση των θεμάτων αυτών. Πρόκειται για, υπάρχει μάλλον συγκεκριμένη υπηρεσία στις ΙΠΑ που ασχολείται με τα ναρκωτικά στο Αφγανιστάν. 13 άτομα αριθμούσε η υπηρεσία αυτή στην αρχή της θητείας του Πρόεδρου Ομπάμα και πλέον ε, αριθμεί 81 μέλη. Αυτό νομίζω ότι είναι ενδεκτικό σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ε, αγροτών στο Αφγανιστάν, θα πρέπει να αναφέρουμε και θέματα του πόσο θυμωμένο είναι το κοινό. Δεν ε, απαντάω ίσως στο ερώτημά σας, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε την στρατηγική μας από άλλη οπτική γωνία, που ελπίζουμε να έχει πιο μεγάλο αντίκτυπο για θέματα επανενσωμάτωσης. Ειλικρινά δεν έχω διαβάσει το άρθρο του στρατηγού Μακρίσταλ σήμερα το πρωί στους Financial Times. Να σας πω όμως ότι οποιαδήποτε διαδικασία επανενσωμάτωσης θα πρέπει να είναι αφγανικής πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να είναι ένα θέμα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και περαιτέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ μόνη μου στην παρούσα φάση. Κύριε Πρέσβη, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια κι εσείς. Εν κατακλείδη. Χαίρομαι που συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση. Ήταν μια Εξαιρετική ευκαιρία για μένα να βοηθήσω, να υποβοηθήσω την υπόθεση του Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι βλέπουμε την κατάσταση με μεγαλύτερη διάβια. Το Αφγανιστάν έχει προδέψει. Ε, ε, εδώ και 8 χρόνια φτάσαμε σε ορισμένα και εκτιμένα και πιστεύω ότι ο αφγανικός λαός με την διεθνή σύνδρομη θα προδεύσει ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια και την στρατιωτική αρρωγή για να βγούμε από αυτή την κρίση που ε, διαρκεί εδώ και 33 χρόνια. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ όλους, λέει ο Πρόεδρος. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για ώρες και μέρες. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μετά τη διάσκεψη του Λονδίνου και υπό το φως των συμπερασμάτων θα δούμε πώς θα προωθήσουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης. Θα έχουμε ευρύτερες ε, συζητήσεις στα πλαίσια της ΑΦΕΤ και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις ειδικέ ε, εξελίξεις στον τομέα ασφαλείας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, ευχαριστώ και τη Γραμματεία και τους διερμηνείς. με ακούλπα εγώ φταίω που ε, καταπατήσαμε το χρόνο σας, αλλά την επόμενη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα τα πούμε την ε, Τετάρτη με την Μάντλεν Ολμπράιτ.